Welcome uh, Σας καλωσορίζουμε. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στην κοινή συνάντηση των Επιτροπών Οικονομικών Υποθέσεων και Κοινωνικών και Απασχόλησης. Θα συζητήσουμε το θέμα των συστάσεων αναχώρα. Έχουμε προσκαλέσει τον κύριο Ντομπρόσκης, Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την κυρία Τάισεν, Επίτροπο για τα θέματα απασχόλησης και κινητικότητας εργασίας και τον Πιερ Μοσκοβισή, υπεύθυνο για θέματα οικονομικά, χρηματοδοτικά, φορολογικά. Θα υπάρξει συμπροεδρία ανάμεσα στις δύο κοινοβουλευτικές επιτροπές και θα ξεκινήσω δίδοντας τον λόγο στον κύριο Ντομπρόσχες να μας κάνει μια σύντομη εισαγωγή. 6-7 λεπτά παρακαλώ, όχι περισσότερο, για να υπάρξει χρόνος και για τους υπόλοιπους ομιλητές και για τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ξεκινώντας να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και την ευκαιρία ανταλλαγής απόψεων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο και πιο συγκεκριμένα για τις ε, αναχώρα ειδικές συστάσεις. Πριν περάσω στο θέμα αυτό, τον CSR δηλαδή, θα ήθελα να πω ότι κάνουμε την συζήτηση αυτή σήμερα μία μέρα μετά από την δημοσίευση της έκθεσης των πέντε προέδρων για την ολοκλήρωση της ε, <clears throat> Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και γι' αυτό θα πρέπει να σταθούμε και λίγο στα θέματα τα οποία έχουν σχέση με το λεγόμενο streamlining και το ευρωπαϊκό εξάμεινο. Η έκθεση είναι θα έλεγα μια ρεαλιστική βάση για την ενίσχυση της νομισματικής ένωσης. Ε, και βασίζεται σε αυτά που μάθαμε πολλές φορές με υψηλό τίμημα για τον τρόπο που λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και στον οικονομικό τομέα και στον πολιτικό και στον χρηματοπιστωτικό. Θα ήθελα τώρα να έλθω σε κάποιες από τις βασικές συστάσεις τις οποίες έχουμε συζητήσει στα πλαίσια της προσπάθειας ολοκλήρωσης της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης. Η ολοκλήρωση αυτή θα πρέπει να συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα με την κοινωνική συνοχή και την σύγκληση. Απαιτείται υψηλότερος διαμοιρασμός κινδύνων ε, και στον τομέα των τραπεζών της ε, Πιστοτικής Ένωσης, ε, των κεφαλαίων και της σταθεροποίησης της λειτουργίας των χρηματοπιστωτικών και θα, και θα πρέπει να υπάρξει επίσης και υψηλότερο επίπεδο διαμοιρασμού κυριαρχίας επί τη βάση φυσικά των ισχύουσων συνθήκων. Θα πρέπει να προθήσουμε την καινοτομία, να προθήσουμε δημοσιονομικές μεταρρυθμίσεις, να εμβαθύνουμε την νομισματική ένωση, να διασφαλίσουμε την επιτυχία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, και τις επόμενες εβδομάδες θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε αυτά πιο αναλυτικά. Έρχομαι τώρα στο θέμα που μας απασχολεί περισσότερο σήμερα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που δίνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να έλθει εδώ και να παρουσιάσει το θέμα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου σε σχέση με τις αναχώρα συστάσεις είναι η πρώτη έκδοση αν θέλετε των συστάσεων αυτών στα, για το νέο σύνολο των επιτρόπων και για το κοινοβούλιο, αυτό το κοινοβούλιο. Όπως ανακοινώθηκε και στην ετήσια αίτηση, έκθεση ανάπτυξης για το 2015 που σας παρουσίασα πριν μερικούς μήνες, εμείς προσπαθούμε να αυξήσουμε την αίσθηση ιδιοκτησίας της μεταρρυθμιστικής διαδικασίας και προώθησης διαφορετικών μεταρρυθμίσεων. Το πρώτο στοιχείο αφορά την ίδια τη διαδικασία. Δημοσιεύθηκαν οι εκθέσεις αυτές τον Φεβρουάριο στα πλαίσια της MIB, της διαδικασίας μακροοικονομικής ανισορροπίας. Έχει προωθηθεί η μελέτη τους λοιπόν σε σχέση με τον προηγούμενο χρόνο. Είναι συστάσεις οι οποίες έχουν σαν στόχο να υπάρξει ένας μεγαλύτερος διάλογος, ένας μεγαλύτερος σε βάθος διάλογο με όλους τους εμπλεκομένους, όχι μόνο τις κυβερνήσεις των κρατών μελών, αλλά και των κοινοβουλίων και των κοινωνικών εταίρων. Στο πλαίσιο αυτό επισκέφτηκα πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συζήτησα τα θέματα αυτά με εκπροσώπους των κυβερνήσεων και των κοινοβουλίων και με την βοήθεια του Πιέρ και της Μαριάν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε αρκετές μορφές πολιτικής συζήτησης. Η αποδοχή των προτάσεών μας ήταν αρκετά θετική, αν και έχουν υπάρξει κάποιες διαφοροποιήσεις και διαφορετικές απόψεις σε συγκεκριμένα στοιχεία. Έρχομαι στο δεύτερο θέμα, το λεγόμενο streamlining, το οποίο ε, μας επιτρέπει να ελέγξουμε τις διαδικασίες καλύτερα αναφερόμαστε στις φετινές αυτές συστάσεις στα κομβικά θέματα στα οποία απαιτείται άμεση δράση από τα κράτη-μέλη. Οι συστάσεις του 2015 ε, υπογραμμίζουν τις ανισότητες τις μακροοικονομικές όπου υπάρχουν. Ας πούμε υπερβολικά ελλείμματα, Βουλγαρία, Κροατία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία. Οι συστάσεις είναι πιο συγκεκριμένες και σφαιρικότερες ταυτόχρονα. Τα CSR αυτά καλύπτονται ε, και προβλέπεται να καλυφθούν σε μία περίοδο από 12 με 18 μήνες. Η προσπάθεια streamlining έχει οδηγήσει σε μια ουσιαστική μείωση του αριθμού των συστάσεων κατά το 1 τρίτο. Η απουσία βέβαια συγκεκριμένων συστάσεων για ένα συγκεκριμένο τομέα δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι θα πρέπει να, σταματήσει η μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Πιο συγκεκριμένα πάλι για το 2015 ε, όπως είπα ασχολούνται οι συστάσεις αυτές με συγκεκριμένους τομείς κατά προτεραιότητα αύξηση παραγωγικότητας, αφαίρεση εμποδίων για την διευκόλυνση των παραγωγικών επενδύσεων, σταδιακές μεταρρυθμίσεις στις υπηρεσίες, στην παραγωγή προϊόντων, για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και δημοσιονομικές πολιτικές υπεύθυνες οι οποίες αποκαθιστούν μια ισορροπία και μια αηφορία ανάμεσα στους βραχυπρόθεσμους διορθωτικούς στόχους και, τις μακροπρόθεσμες, και τους μακροπρόθεσμους. Θα πρέπει τα μέτρα τα κυβερνητικά αυτά, οικονομικά τα οποία λαμβάνονται να έχουν σαν βασικό στόχο την στήριξη της ανάπτυξης και της διευκόλυνση επίσης του κοινωνικού διαλόγου. Για το σύνολο αναφέρομαι της περιοχής του ευρώ. Πρέπει να βελτιωθεί φυσικά περαιτέρω η οικονομική διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης και συμπερασματικά θα έλεγα ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει σαν στόχο την συνολική αντιμετώπιση των οικονομικών προβλημάτων όπως αυτά έχουν εντοπιστεί μέχρι τώρα και γι' αυτό οι χώρες συνεργάζονται με αποτελεσματικό τρόπο, αυτό διαπιστώνουμε μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε τη συνεργασία μαζί τους ε, σε στενότερο επίπεδο. Ε, αυτή η προσπάθεια την οποία κάνουμε για πιο επικεντρωμένο ευρωπαϊκό εξάμεινο και για την αύξηση του λεγόμενου streamlining στο εξάμεινο θα το καταστήσουν πιο ελκυστικό. Ευχαριστώ. Η κυρία Τάισεν έχει το λόγο, η υπεύθυνη επίτροπος για την κινητικότητα των εργαζομένων και την απασχόληση. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Αγαπητοί Πρόεδρε, αγαπητά μέλη των Επιτροπών, θα ήθελα να επικεντρωθώ στι συστάσει για την απασχόληση από πλευρά τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή προ τα κράτη-μέλη. Από ό,τι ξέρετε, αποτελούν ένα σημαντικό τμήμα τη άσκηση για το Ευρωπαϊκό Εξήμενο. Ξέρετε ότι το ποσοστό τη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει μειωθεί στο 9,7% τον περσινό Απρίλιο το πιο χαμηλό ποσοστό από το Σεπτέμβριο του 2011 και παρά το γεγονός ότι στην Ευρωζώνη εξακολουθεί να είναι σε αντιψήφια επίπεδα η ανεργία στο 11,1% ως τώρα τα ποσοστά αυτά μειώνονται. Ωστόσο είναι πάρα πολλές οι προκλήσεις που έχουμε ενώπιόν μας καθώς όπως ξέρετε έχουμε ακόμα 23,5 εκατομμύρια ε, ανέργους στην Ευρώπη και 4,6 εκατομμύρια εξ αυτών είναι νέοι. Με μεγάλες αποκλήσεις μεταξύ των κρατών μελών. Στην παρούσα φάση μπορούμε να δείξουμε μια νέα εμπιστοσύνη στην Ευρωζώνη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χαλαρώσουμε και να εφησυχαστούμε. Θα πρέπει να ε, επιταχύνουμε την ανάκαμψη προκειμένου να δώσουμε μια καινούργια πνοή στην αγορά εργασία μας ε, προκειμένου να μην ε, μένει κανείς στο μέλλον πίσω. Οι συστάσεις για την απασχόληση λοιπόν ε, εστιάζονται στις πιο βασικές μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας και στο πώς μπορούν να ενταχθούν αυτοί που έχουν χτυπηθεί πιο φαναρά από την κρίση. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η ανεργία των νέων και η μακροπρόθεσμα άνεργη. Σε ό,τι αφορά την νεολαία, έχουμε ξεκινήσει να βλέπουμε τα πρώτα αποτελέσματα. Πολλά άτομα τα οποία μεταξύ του Μαρτίου του 2014 και του Μαρτίου του 2015 έχουν βρει ε, δουλειά. Αλλά ένα στους πέντε στην αγορά εργασία εξακολουθούν να είναι χωρίς, ε, δουλειά και πιο πολύ, η μισή σχεδόν από τις 23,5 εκατομμύρια ανέργους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι μακροπρόθεσμα άνεργοι. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις ε, επίσημα στοιχεία για την ε, ανεργία και να συνεργαστούμε με τις αναλόγες υπηρεσίες. Εστιαζόμαστε σε στοχευμένα μέτρα για να αυξήσουμε τη συμμετοχή στην αγορά εργασίας για τις ευάρετες ομάδες όπως τις ε, γυναίκες, τους ηλικιωμένους, τους μετανάστες. Η βελτίωση των ικανοτήτων και η εκπαίδευση αποτελεί, αποτελούν ένα κλειδί. Παράγοντα κλειδί για την απασχολησιμότητα και την πρόσβαση στην αγορά εργασία και οι βασικέ μεταρρυθμίσει που απαιτούνται συμπεριλαμβάνουν την πρόληψη τη εγκατάλειψης του σχολείου, διαβιομάθηση, πρόσβαση στην εκπαίδευση για τι ευάλωτε ομάδε και μεταρρύθμιση τη ε, ε, εκπαίδευσης. Σε ό,τι αφορά τους μισθούς θα πρέπει να λάβουμε υπόψη τα επίπεδα παραγωγικότητας και εδώ να βρούμε μια ισορροπία μεταξύ ανταγωνιστικότητας, ε, δημιουργίας θέσης εργασίας και ε, ζήτησης. Και εδώ πέρα λοιπόν αναγνωρίζεται η αξία και των ε, κοινωνικών φορέων. Οι παρεκκλήσεις στις τάσεις για την ένδυα έχουν, αρχίσει, έχουν συνεχίσει να αυξάνονται τα κράτη-μέλη λόγω της αύξησης της ένδυας στις χώρες της Ευρωζώνης που έχουν χτυπηθεί πιο έντονα από την κρίση. Οι συστάσεις οι φετινές εστιάζονται στη μείωση της ένδυας και της κοινωνικού αποκλεισμού πληρώνοντας τα χάσματα στο δίκτυο, το κοινωνικό ιστό και στο δίκτυο ασφαλείας των κρατών μελών. Επίσης δίνεται μεγαλύτερη προσοχή στη φύλαξη των παιδιών και την ε, έγκαιρη προσχολική εκπαίδευση για τα παιδιά από πιο μειονεκτούντα περιβάλλοντα. Ιδιαίτερα ε, εστιαζόμαστε και στις ε, χώρες με μεγάλο πληθυσμό Ρωμά. Εστιαζόμαστε στην ενίσχυση της βιωσιμότητας και της καταλληλότητας με την διασφάλεια, διασφάλιση μιας μακρύτερης καριέρας, ε, μειώνοντας τις δυνατότητες προώρης ε, συνταξιοδότησης, βελτιώνοντας την αποσχολησιμότητα των πιο ηλικιωμένων και ε, την αποσχολησιμότητα ανδρών και γυναικών. Τέλος, σε ό,τι αφορά τα θέματα της υγείας και της υγειονομικής περίθαλψης, ένας μεγάλος τομέας της οικονομίας που δεν έχουμε ακόμα καταφέρει να ελέγξουμε, αλλά όπως ξέρετε η υγειονομική περίθαλψη διασφαλίζει ότι όλοι έχουν πρόσβαση στα, στις υπηρεσίες ε, υγείας, όχι μόνο οι πιο πλούσιοι. Άρα τα βασικά μηνύματα για την ε, υγειονομική περιθάλψη είναι η αποδοτικότητα βάση κόστου ε, και η παραγωγικότητα, η αποδοτικότητα. Και για να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε, πρέπει να πούμε συνοψίζοντας ότι έχει έρθει το πλήρωμα του χρόνου για μια μεταρρύθμιση στην Ευρώπη που χρειάζονται, πρέπει να καταφέρουμε να δούμε πέρα από τα καταπήγοντα ζητήματα που ανακύπτουν κατά την κρίση και να δούμε τι χρειάζεται για μεγάλη αποδοτικότητα προκειμένου να δοθεί και μια μεγάλη όθηση στην ανταγωνιστικότητά μας σε παγκόσμιο προσκήνιο γιατί εκ παραλλήλου θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να ενισχύσουμε το ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Η Ευρωπαϊκή μας ε, Επιτροπή πιστεύει ότι με το νέο συντονισμένο μοντέλο, εναρμονισμένο μοντέλο, μπορούμε να δώσουμε τις προτεραιότητες εκεί που χρειάζεται και έχουμε κάνει το όσο μας αναλογούν. Τώρα πλέον επαφή στα μέλη να φροντίσουμε την εφαρμογή. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Πιέρ Μοσκοβισή, Επίτροπο για Οικονομικά Ζητήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι ευρωβουλευτές, αγαπητοί συνάδελφοι. Οι θετινές συστάσεις καλύπτουν τις κύριες προτεραιότητες οικονομικές και κοινωνικές που απαιτούν τα κράτη-μέλη να προσέξουν τους επόμενους 12 με 18 μήνες. Καλύπτουν διάφορες προτεραιότητες. Πολλές συστάσεις έχουν σαν στόχο να διορθώσουν τις ανισορροπίες που υπάρχουν στο δημοσιονομικό τομέα. Ε, βλέπουμε ότι υπάρχουν προβλήματα στις επενδύσεις. Γι' αυτό και θέλουμε να βελτιωθεί το κλίμα υπέρ των επενδύσεων. Άλλη σύσταση αναφέρεται στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, με συγκεκριμένες συστάσεις για τις χώρες εκείνες που έχουν υπερβολικές ανισορροπίες. Οι μισές χώρες μέλη καλούνται ακόμα να κάνουν περισσότερες μεταρρυθμίσεις στο συνταξιδοτικό του σύστημα, με διαφορές βέβαια και αποχρώσεις ανάλογα με την ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας. Στον τομέα των δημοσιοοικονομικών, οικονομικών, όλες οι χώρες μέλη εκτός από 9 αποτελούν αντικείμενο σύσταση. Δανία, Εστονία, η Φιλανδία, η Μάλτα, Κατοχώρες, η Ρουμανία η Σουηδία, η Σλοβενία και η Σλοβακία. Οι άλλες 17 καλούνται να πάρουν ειδικά μέτρα να μειώσουν, για παράδειγμα, τη δημοσιονομική πίεση επί της εργασίας και να διευρύνουν τη φορολογική τους βάση. 17 και 9 ναι, θα μου πείτε κάνει 26. Ε, δεν μιλάω για την Κύπρο και την Ελλάδα, οι οποίες όπως γνωρίζετε είναι δύο χώρε που βρίσκονται υπό πρόγραμμα. Τέλος, Κάνουμε και συστάσεις ειδικέ για την ε, δημοσιονομική πολιτική και την οικονομική διακυβέρνηση για όλες τις χώρες πλην 7. Σουηδία, Λουξεμβούργο, Γερμανία, Κατοχώρες και Σλοβακία. Και γιατί, γιατί χώρες αυτές συνάδουν με το Σύμφωνο Σταθερότητα και Ανάπτυξη, συνεπώ δεν κάναμε δημοσιονομικέ συστάσει για αυτέ και επαναλαμβάνω ότι η Ελλάδα και η Κύπρο αποτελούν μια χωριστή κατηγορία γιατί βρίσκονται υπό πρόγραμμα. Οι δημοσιονομικέ συστάσει σκοπεύουν να διασφαλίσουν ότι όλε οι χώρε ε, δουλεύουν σύμφωνα με το Σύμφωνο σταθερότητα και ανάπτυξη ή μπορούν να βελτιώσουν τη διακυβέρνησή του σε διάφορα επίπεδα. Επιτρέψτε μου να πω περισσότερο σε βάθο όσον αφορά τη δημοσιονομική πολιτική. Το δημοσιονομικό προφίλ στην Ευρώπη πρέπει να ξέρετε ότι βελτιώνεται. Οι περισσότερε χώρε μέλη έχουν μειώσει τα ελλείμματά τους. Το 2014 το συνολικό έλλειμμα των κυβερνήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση έπεσε κάτω από το 3% του ΕΠ για πρώτη φορά από το 2008 και το έλλειμμα στην Ευρωζώνη ε, μειώθηκε στο 2,4% και πιστεύουμε ότι η τάση αυτή θα συνεχιστεί και το 2015 και την επόμενη χρονιά. Για πρώτη φορά το, η σχέση του χρέους με το ΕΠ βελτιώνεται φέτος. Πολύ σημαντικό αυτό. Συγχρόνως διαπιστώνουμε ότι οι περισσότερες ε, χώρες που δεν τα κατάφεραν, δεν πέτυχαν το στόχο του ελλείμματος, οι μισές από αυτές περίπου προβλέπεται να αποκλίνουν από τις απαιτήσεις του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης φέτος. Οι περισσότερες από τις χώρες μέλη δεν προβλέπεται να συμμορφωθούν με το σύμφωνο, ούτε το 2016, έξι χώρες στο προληπτικό σκέλος, που κινδυνεύουν δηλαδή να αποκλίνουν σημαντικά, και κάποιες άλλες στο διορθωτικό σκέλος, που ίσως δεν θα μπορέσουν ή τουλάχιστον δεν είναι σίγουρο ότι θα μπορέσουν να κάνουν τις διορθώσεις που χρειάζεται έγκαιρα. Η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία και η Γαλλία δηλαδή. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό οι χώρες μέλη να υποφεληθούν από τη σημερινή περίοδο χαμηλών επιτοκίων και ευκαιριών που προσφέρονται και να συνεχίσουν την πολιτική τους μείωσης των ελλημάτων και του χρέους τους. Κροατία ήθελα να πω, όχι Ουγγαρία. Βλέπετε εδώ έβλεπα HR και μπερδεύτηκα. Ενώ λοιπόν οι χώρες μέλη έχουν ε, δημοσιονομικά, κάποια δημοσιονομικά πλεονεκτήματα, αυτές πρέπει να δώσουν νέα όθηση στις επενδύσει τους. Η Γερμανία για παράδειγμα, αλλά όλες πρέπει να συνεχίσουν να φροντίζουν για τη βιωσιμότητα των δημοσιονομικών τους. Επιτρέψτε μου τώρα να περάσω στις προτάσει μα Για τη Μάλτα και την Πολωνία προτείνουμε να κλείσουμε τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματο, γιατί η Μάλτα έχει κατεβάσει το έλλειμμά της κάτω από το 3% του ΑΕΠ με βιώσιμο τρόπο και ε, άρα συμμορφώνεται με τους κανόνες για το χρέος από το 2014. Για την Πολωνία υπήρχαν διάφορα περίπλοκα μέτρα, έγινε μεταρρύθμιση του συνταξιδοτικού τους, τώρα όμως βρίσκεται κάτω από το 3% και αυτή, οπότε το ίδιο ακριβώς προτείνουμε και για την Πολωνία. Όμως λέμε ότι δεν πρέπει να αντιστραφεί η μεταρρύθμιση που έγινε στο συνταξιδοτικό. Για το Ηνωμένο Βασίλειο τώρα δεν διόρθωσε το υπερβολικό έλλειμμα και στην προθεσμία που πρότεινε το Συμβούλιο, γι' αυτό και προτείνονται νέε αποφάσει με νέα προθεσμία για τα έτη 2016 και 2017. Για τη Φιλανδία στις 13 Μαΐου εκδώσαμε έκθεση με την οποία αξιολογούμε την παραβίαση των κριτηρίων του χρέους και του ελλείμματος λέγοντα ότι δεν υπάρχει συμμόρφωση με αυτά τα δύο κριτήρια. Έκτοτε βέβαια έχουμε νέες πληροφορίες από την κυβέρνηση. Το κυβερνητικό πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορα μέτρα εξυγένσης για το 2016 μέχρι το 2019. Επιπλέον προβλέπονται και διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν δεν θα προτείνει τίποτα νεότερο, θα παρακολουθήσει την κατάσταση και θα συνεχίσει το διάλογο με την κυβέρνηση προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες απαντήσεις. Η Γαλλία στις 10 Ιουνίου παρουσίασε έκθεση με μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί στις συστάσεις του Συμβουλίου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το εξετάζει και θα πει πολύ σύντομα ποια είναι η κατάσταση. Βλέπουμε ότι τα πράγματα πάνε προς τη σωστή κατεύθυνση, παρόλο που πολλά μένουν ακόμα να γίνουν συγκεκριμένα. Τέλος. Όσον αφορά τη διαδικασία μακροοικονομικών ανισορροπιών, εξετάζουμε τα εθνικά προγράμματα μεταρρύθμισης βλέπουμε ότι είναι φιλόδοξα και λεπτομερή. Και γι' αυτό δεν έχουμε προτείνει ε, καμιά διαδικασία ε, μέχρι το Μάρτιο για καμία χώρα. Γιατί θέλουμε να βοηθήσουμε τις χώρες και να τις στηρίξουμε στην ανάκαμψή τους. Βέβαια, κάποιες χώρες πρέπει να κάνουν παραπάνω προσπάθειες για να ξεπεράσουν τις ανισορροπίες που υπάρχουν στα δημοσιονομικά τους. Πάντω, η οικονομική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπή επιβεβαιώνεται. Η Ευρώπη πρέπει να επιταχύνει τις διαστατικές μεταρρυθμίσει και πρέπει να υπογραμμίσει ακόμα περισσότερο τις επενδύσεις, προχωρώντας βέβαια και με υπευθυνότητα στην εξέλιξη των ε, δημοσίων οικονομικών. Ο κύριος στόχος τους επόμενους μήνες είναι να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας προκειμένου να εφαρμοστούν οι συστάσεις μας. Αυτές τις τελευταίες εβδομάδες μάλιστα επισκέφθηκα πολλές χώρες μέλη για να παρουσιάσω και να εξηγήσω τις συστάσεις μας και είμαι πεπισμένος ότι οι προσπάθειες αυτές βελτιώνουν την κατανόηση και σε εθνικό επίπεδο. Γιατί όπως είπαμε πρέπει ο κόσμος να ενστερνίζεται. Οι χώρες, το κοινοβούλια, η κοινή γνώμη, οι οικονομικοί και οι κοινωνικοί φορείς πρέπει να ενστερνίζονται. Τις καταλαβαίνω αυτές τις συστάσεις και να τις σκοπιούνται. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας εξαίρετος εταίρος προκειμένου να στηρίξει την προσπάθειά μας αυτή. Γι' αυτό και έχουμε αυτήν την από κοινού ακρόαση σήμερα. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, με δύο λόγια αυτές είναι οι λεπτομέρειες των προτάσεών μας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Μοσχοβησή. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κύριε Τόμας Χέντελ. Αν θέλετε κι εσείς να πείτε κάποια πράγματα στα μέλη της Επιτροπής Απασχόλησης τουλάχιστον, κύριο Χέντελ. Χαίρομαι που βρίσκομαι με μεγάλη παρέμβαση εδώ και θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι μου έστειλαν ευχές κατά τη διάρκεια της ασθενειάς μου. Θα ήθελα να σας πω ότι θα μου χρειαστεί κάποιος χρόνος για να ξαναμπω μέσα στα πράγματα, αλλά κάνω ό,τι μπορώ και υπολογίζω στην υποστηριξή Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους αντικαταστάτες μου στην Μαρίτα Ιουσκόκ, η οποία κατά τους 11 μήνες αυτούς αναγκάστηκε να κάνει μεγάλο τμήμα της δουλειάς όλα όσα άφησα πίσω μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Μαρίτα λοιπόν. Ελπίζω να έχω την υποστήριξή σου και τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό ήταν κάτι το ε, ιδιαίτερο για μένα. Επανέρχομαι λοιπόν στην ε, καθημερινότητα. Θα δώσω το λόγο σε μια πρώτη φάση τουλάχιστον, σε μια σειρά από μιλητές, το, το συντομότερο βέβαια δυνατό για τον καθένα, τρία λεπτά οι συγητές για την έκθεση για το εξάμεινο. Ποιος αντικαθιστά τον εισηγητή. Έχετε το λόγο. Μην ανησυχείτε, μόνο για σήμερα λέει η κυρία Χιούμπνερ. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι στρέφομαι προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Έχετε καταστήσει ευτυχή τον κύριο Ροζάτη. Καταρχάς, έχετε συγκεντρώσει την προσοχή σας στα τρία βασικά σημεία των συστάσεων αναφόρα. Έχετε εντοπίσει σωστά τους παράγοντες οι οποίοι καθιστούν εύθραυστη την ανάπτυξη και επίσης η αναφορά σας για τον μηχανισμό ευελιξίας είναι κάτι το ιδιαίτερα θετικό. Έχει κάποιες ερωτήσεις. Λοιπόν, πρώτον, δεν είναι ξεκάθαρο με ποιο τρόπο θέλει να δώσει κίνητρα στα κράτη-μέλη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έτσι ώστε να τα να εφαρμόσουν τις συστάσεις. Δεύτερον τώρα για την έκθεση των πέντε προέδρων για την κινητοποίηση των κρατών μελών να συνεχίσουν με διαρθρωτικές αλλαγές καθοριστικές για τη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Και τρίτον για τις μικρομεσαίες. Έχουμε ήδη συζητήσει για τις μικρομεσαίες υπάρχει ανάγκη για τη βελτίωση της χρηματοδότησης της μικρομεσές και πώς έχουμε κάνει βήματα στην πρόσβασή τους σε χρηματοδότηση. Μία συμπληρωματική ερώτηση. Οι συστάσεις αυτές για την Ευρωζώνη, ποιος είναι αυτός ο οποίος ε, θα εφαρμόσει αυτά τα οποία προτείνεται για το σύνολο της Ευρωζώνης όπως κάνετε τις συστάσεις σας. Νομίζω θα δώσουμε το λόγο επίσης στον εισηγητή της Επιτροπής Απασχόλησης, τον Πριέτο. Κύριε Πριέτο, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και τους Επιτρόπους για τις παρεμβάσεις τους σε αυτήν τη μεικτή Επιτροπή. Είναι σαφές ότι οι συγκεκριμένες αυτές στάσεις συνολικά παραπέμπουν σε καλές προθέσεις, σε κάποιες βασικές αρχές και απαιτείται να καθορίσουμε σωστότερα την πολιτική των κρατών μελών για τα επόμενα θα έλεγα χρόνια είναι καθοριστική. Το θέμα είναι βέβαια να δούμε και σε ένα επίπεδο αρκετά πιο λεπτομερές τι ακριβώς χρειάζεται να γίνει. Το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζει η Ευρώπη σήμερα, συνάδελφοι, είναι το πρόβλημα της ανισότητας. Α, πολλοί διεθνείς οργανισμοί λέγουν ότι η ανισότητα αυτή δημιουργεί οικονομικά προβλήματα, επιβραδύνει την ανάπτυξη και δημιουργεί επίσης προβλήματα εις βάρος της κοινωνικής συνοχής. Υπάρχει μια αντιστρόφως ανάλογη σχέση ανάμεσα στις αποδόσεις τις οποίες ε, έχουν οι επενδύσεις στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Η διαφορά ανάμεσα στο φτωχότερο 10% και στο ψηλότερο και πλουσιότερο 10% έχει πολλαπλασιαστεί. Λοιπόν, το θέμα είναι αν μπορούμε να μειώσουμε αυτή την ανισότητα, ανισότητα η οποία περιέχει θα έλεγα τρία βασικά χαρακτηριστικά. Το πρώτο είναι η φορολογία. Η φορολογία είναι πάρα πολύ άνηση και άδικη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φορολογεί την εργασία περισσότερο από το κεφάλαιο. Είναι σαν παράδειγμα υψηλή φορολογία στις χαμηλές αμοιβέ, στους χαμηλούς μισθούς και η φορολογία αυτή συν της άλλης δεν είναι και αναδιανεμητική. Λοιπόν, και με τους δείκτες τους οποίους χρησιμοποιούμε φοβάμαι ότι δεν μπορούμε να έχουμε και μια ξεκάθαρη εικόνα για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα και γι' αυτό χειροτερεύουν οι συνθήκες χρηματοδότησης σε τομείς όπως η εκπαίδευση και κυρίως η υγεία και φυσικά υπάρχει η τρομερή αύξηση της μακροπρόθεσμης ε, ανεργίας. Το θέμα της ε, μεταρρύθμισης ε, της αγοράς εργασίας. Είχε πει η κυρία Μέρκελ ότι θα πρέπει να υπάρξει μια μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά εργασίας της χώρας της βέβαια και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Υπάρχει αυτή η ευελιξία. Αυτό σημαίνει ότι το 40% των εργαζομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι με επιμέρους ε, συμβάσεις οι οποίες είναι περιορισμένου χρόνου και οδηγούν στην ε, αμοιβή των εργαζομένων με πολύ χαμηλούς μισθούς και τους οδηγούν στη φτώχεια παρότι εργάζονται. Οι προτάσεις λοιπόν της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν ότι μία αύξηση έστω και κατά 1% των μισθών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των εργαζομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα καταστήσουν, λέγει, μη ανταγωνιστική την ευρωπαϊκή οικονομία. Αυτό είναι λάθος. Υπάρχει ύφεση και η ύφεση οδηγεί στην ανισότητα και στις τρομερές διαφορές απαιτείται μια αύξηση των μισθών, αυτό θα δώσει ενέργεια στην ευρωπαϊκή οικονομία και θα αποκαταστήσει την ισότητα ανάμεσα στους εργαζομένους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα, έτσι θα ζήσει το κοινωνικό μας πρότυπο. Θα δώσω το λόγο για να απαντήσει ο κύριος Ντομπρόσκης πρώτος. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες πρώτες απαντήσεις, ίσως και οι υπόλοιποι επίτροποι. Για τους βασικούς στόχους, τους κεντρικούς στόχους ε, που έχουν οι συστάσεις αυτή τη φορά αναχώρα. Σας ευχαριστώ καταρχάς για τα θετικά σας λόγια. Τώρα για την εφαρμογή αυτών των συστάσεων. Το θέμα αυτό είναι βέβαια η εφαρμογή τους. Αυτό το υπογραμμίζουμε συνεχώς. Η ερώτηση μας τίθεται συνεχώς. Είναι συστάσεις κύριοι, δεν είναι διαταγές αυτές, αυτές οι προσπάθειες που κάνουμε. Απαιτείται να καταστήσουμε τους εμπλεκομένους να νιώθουν ότι ελέγχουν οι ίδιοι, ότι είναι δικές τους οι διαδικασίες αυτές να προωθήσουμε έτσι ακόμα περισσότερο τη διαδικασία αυτή των συστάσεων προκαλώντας συζητήσεις, προκαλώντας επιστροφή ενημέρωσης από τα κράτη-μέλη και να καταλήγουμε κάθε φορά σε ισόρροπες τέτοιες συστάσεις κατανοητές από τα κράτη-μέλη και εφαρμόσιμες. Τώρα για τις συστάσεις προς την περιοχή του ευρώ, για την ευρωζώνη. Ε, σε επίσημο επίπεδο απευθύνονται σε αυτό που ονομάζουμε Eurogroup και θα πρέπει το Eurogroup σαν σώμα να συζητήσει συνολικά, σαν συλλογικό όργανο καλύτερα, να συζητήσει τον τρόπο με τον οποίο θα συντονίσει καλύτερα τις ευρωπαϊκές χώρες και τις πολιτικές της Ευρωζώνης έτσι ώστε να εφαρμόσει σωστά τις συστάσεις αυτές. Κάποια άλλα στοιχεία για την ανισότητα των εισοδημάτων. Εδώ η κυρία Τίσεν ίσως έχει να προσθέσει κάποια πράγματα και για τα θέματα της φορολογίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία, την λεγόμενη πρωτοβουλία της δίκαιης φορολογίας και για, τον επιχειρηματικό, για την ε, φορολογία των επιχειρήσεων. Νομίζω ότι εδώ ο Πιέρ μπορεί να προσθέσει κάποια στοιχεία ενδιαφέροντα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τάισεν τώρα έχει το λόγο. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε. Θα χρησιμοποιήσω τους δερμηνείς και θα απαντήσω στη γλώσσα μου. Θα ήθελα λοιπόν καταρχάς ε, να απαντήσω στην ερώτηση του κυρίου Κουτιέρες Πέτο. Η μελέτη, η έρευνα του Διεθνές Νομισματικού Ταμείου για την ανισότητα που αυξάνεται. Για το γεγονός ότι αυτή η αυξούμενη ανισότητα αποτελεί ένα εμπόδιο στην ανάπτυξη. Αυτό επιβεβαιώθηκε και μάλιστα είχε προηγηθεί και μία ε, έρευνα του ΑΣΑ που καταδεικνύει ότι αυξάνεται ακριβώς αυτό το, αυτή η ψαλίδα της ανισότητας και ότι αυτό αποτελεί ένα πρόσκομα για την ανάπτυξη των χωρών και ότι θα πρέπει να υπάρξει ανακατανομή είτε μέσω κοινωνικών ε, μέσων είτε μέσω των, ε, της προκειμένου να, υπάρχει, να υπάρξει ανάπτυξη και να μην ε, ανακόπτεται αυτή η ανάπτυξη. Αυτό βέβαια πρέπει να το πετύχουμε με τα μέσα που έχουμε. Θα πρέπει να πείσουμε τα κάτι μελη να λάβουν δράση. Μπορούμε να λάβουμε κι εμείς κάποια μέτρα. Το κάνουμε άλλωστε αυτό με τη συνεργασία κυρίως μεταξύ ημών, με την καλύτερη επιδίωξη των στόχων μας. Θα δείτε λοιπόν και θα διαπιστώσετε ότι στις διάφορες συστάσεις ανά χώρα περιλαμβάνονται συστάσεις σε ό,τι αφορά την συμπερίληψη των πιο ευάλωτων ομάδων και τα μέσα τα οποία θα συμβάλλουν στην άμβληση των ανισοτήτων και στην πρόληψη της περαιτέρω του περαιτέρω κατακαιρματισμού της αγοράς εργασίας υπάρχουν και κάποιες συγκεκριμένε συστάσεις ανά χώρα για το μίσο που πιστεύουμε ότι δεν είναι οι εξελίξεις. Ε, εν γέννη, πρέπει να πετύχουμε μεγαλύτερη σύγκληση. Αυτό το συζητήσαμε και σε μια πρώτη αναγνωριστική συζήτηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αυτό πρέπει να το πετύχουμε με τα μέσα τα οποία έχουμε ήδη στη διάθεσή μας. Πιο πολύ σύγκληση λοιπόν, σύγκληση προς τα πάνω. Γιατί σκοπός είναι να βελτιώσουμε την κατάσταση για τους πολίτες με τα μέσα που έχει στη διάθεση, στη διάθεση της Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέθοδο συντονισμού, συνομιλία, διάλογοι, ε, ορισμός ε, στόχων, ε, αξιολογήσεις από μοντίμους, όλα όσα κάνουμε στα πλαίσια του εξαμήνου, προκειμένου να δοθούν ε, κίνητρα με τα μέσα και τα χρηματοδοτικά κονδύλια τα οποία ήδη διαθέτουμε. Αλλά πιστεύω ότι αυτό αποτυπώνεται και στις συστάσεις αναχώρα, αν τις αναλύσετε σωστά. Άρα θεωρώ ότι μπορούμε να πούμε ότι οι συστάσεις αναχώρα ε, δίνουν μια σαφή κοινωνική σφραγίδα και στο Ευρωπαϊκό Εξάμεινο της φετινής χρονιάς. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μοσκοβίση λέει τώρα η Πρόεδρος. Έχει το λόγο. Όπως το εξήγησα για τις συστάσεις, υπάρχουν 17 χώρες που αποτελούν αντικείμενο συστάσεων όσον αφορά τα δημοσιονομικά τους με δύο στόχους. Να μειωθεί το κόστος της εργασίας και να διαβρύνει τη φορολογική τους βάση. Αλλά όπως που ζήτησε και ο Βαλτής, θα σας πω ποια είναι τα βήματα που κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα δράσης της για την φορολογία. Θα τα παρουσιάσω εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, γιατί στην πραγματικότητα πρόκειται για τη δικιά μας απάντηση σε αυτό που μας ζήτησε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχουν τέσσερις άξονες λοιπόν. Ξεκινάμε από μια βασική ανάλυση που λέει ότι η φορολογία στις επιχειρήσεις δεν ανταποκρίνεται στη σημερινή οικονομία. Φτιάχτηκε για την οικονομία το δεκαετίας του 30 και όχι για τις άιλες ε, και άλλες περίπλοκες μορφές ε, οικονομίας που έχουμε σήμερα. Άρα λοιπόν πρέπει να προσαρμοστούμε στο 21ο αιώνα. Έτσι θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και τις ανισότητες από τις οποίες υποφέρουν συχνά οι φορολογούμενοι και θα μπορέσουμε να αποφύγουμε αυτό το άδειασμα των ταμείων. Γιατί σήμερα υπάρχει μια φοροαποφυγή αποφυγή, φοροδιαφυγή και έτσι δεν γεμίζουν τα ταμεία. Επιχειρήσεις δεν πληρώνουν φόρους και έτσι μειώνεται ο πλούτος. Θα φροντίσουμε να ακολουθήσουμε το CCTB. Είναι κάτι που γνωρίζει πολύ καλά η Μαριάν. Σε δύο φάσεις με μια κοινή βάση καταρχήν και μετά θα προχωρήσουμε επιμέρους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο φαντάζομαι ότι θέλει περισσότερα και εμείς εξάλλου. Αλλά τα τελευταία πέντε χρόνια είχαμε βρεθεί σε διέξοδο. Τώρα λοιπόν προχωράμε σιγά σιγά. Ο δεύτερος άξονας είναι η πραγματική φορολόγηση. Δεν θέλουμε πλέον να δεχόμαστε οι χώρες οι οποίες παράγουν δεν πληρώνουν ή πληρώνουν πολύ λίγους φόρους. Μια πραγματική φορολόγηση σημαίνει ότι πληρώνουμε ε, φορολογία εκεί που παράγεται το αγαθό με τις διάφορες δίτες που μπορεί να προβλεφθούν γι' αυτό. Τρίτος άξονας. Πάντα για τον ίδιο λόγο πιέζουμε υπέρ της διαφάνειας. Είναι η πρώτη πρόταση για οδηγία όσον αφορά την ανταλλαγή πληροφοριών online με το country by country reporting. Στην αρχή θα γίνει μελέτη αντιτύπου, στη συνέχεια διαβούλευση με το κοινό, όχι για να θαυτεί η προσπάθεια, αλλά για να καταστεί συμβατή η διαφάνεια με το πρόγραμμα των επιχειρήσεων. Χρειαζόμαστε και τη στήριξη των επιχειρήσεων. Και τέταρτον, για πρώτη φορά, και το κρίνω και από τα γράμματα που μου φτάνουν, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καταρτήσει κατάλογο με χώρες ή με δάφη που δεν συνεργάζονται προς αυτό το σκοπό. Για να προχωρήσουμε στο name and shame. Κάποιοι προσπαθούν να με πείσουν ότι δεν είναι αλήθεια πως δεν συνεργάζονται. Ωραία, τόσο το καλύτερο να με πείσουν. Αν μία ή άλλη χώρα που βρίσκεται στο κατάλογο αυτό τελικά συμμορφώνεται, τόσο το καλύτερο. Αυτός είναι και ο στόχος του καταλόγου, αν θέλετε, ακριβώς, ώστε οι χώρες να βγουν από αυτό το κατάλογο. Σιγά σιγά. Έχουμε χρησιμοποιήσει τους εθνικούς καταλόγους και έχουμε κάνει μια σύνθεση των καταλογών αυτών. Κάποια χώρα που συμπεριλαμβάνεται σε 10 εθνικούς καταλόγους ε, είναι και σε εμά προτεραιότητα, όπως καταλαβαίνετε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ κύριε Μοσχοβησή. Έχουν ζητήσει διάφοροι από εσά το λόγο. Δεν ξέρουμε κατά πόσο θα υπάρχει χρόνος για κάτι Αν όμω υπάρχει χρόνος, να ξέρετε ότι σας έχουμε σημειώσει στον κατάλογο των ομιλητών. Τώρα, θα δώσω την προεδρία στον κύριο Γκουαλτιέρη. Εσείς αναλαμβάνετε το δεύτερο γύρο της συζήτηση αυτή. Σα ευχαριστώ. Μαρίτα. Θα ξεκινήσουμε με τους σκιώδεις εισηγητές. Ο πρώτος, ο εκπρόσωπος των σκιωδών για 1,5 λεπτό ο καθένας, ο κύριος Σαντ. Να ξεκινήσω συγχαίροντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον τρόπο με τον οποίο προχώρησε στο streamlining του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου προσπαθώντας να συγκεντρώσει τους στόχους. Λέγει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επιστρέφει η ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά ότι οι εξελίξεις που το έχουν βοηθήσει αυτό είναι βραχυπρόθεσμες. Αυτά τα λέει και το IMF, ότι η ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη είναι εύθραστη και γενικά το θέμα είναι και η σχέση με την αγορά εργασίας. Βλέπουμε ότι η κατάσταση ανάκαμψης η σημερινή είναι πάρα πολύ εύθραυστη και οι διαφθρωτικές αλλαγές που θα οδηγήσει στην ευελιξία στις, στις αγορές απασχόλησης έχει τεράστιες κοινωνικές επιπτώσεις. Έχει προκαλέσει ανασφάλεια, έχει προκαλέσει ύφεση, ιδιαίτερα στους νέους, έχει αυξήσει την ανεργία τους και το τι κάνουμε σήμερα δεν θα πρέπει να το αποφασίσουν από μόνες τους οι αγορές. Ε, δείχνουν τα αποτελέσματα των εκλογών στην Δανία, στην Γαλλία και στην Ιταλία ότι επηρεάζεται η ψήφος και από τις οικονομικές εξελίξεις και δυστυχώς πάρα πολλοί πολίτες έχουν αρχίσει να νιώθουν ότι μένουν πίσω και σε επίπεδο γεωγραφικό και σε επίπεδο κοινωνικό στην πρόσβαση στην αγορά εργασίας που για κάποιες περιοχές είναι μακράν του κοινοτικού μέσου όρου. Υπάρχει σύγχυση στον τομέα της σύγκλησης της οικονομικής πολιτικής με μέτρα τα οποία έχουν σαν αποκλειστικό στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας. Δεν μπορούμε εμείς να αφήσουμε στους πολίτες την εντύπωση ότι αντί να διαχειριζόμαστε στην Ευρώπη την αγορά, η αγορά διαχειρίζεται την Ευρώπη. Λοιπόν, θα πρέπει να μην είμαστε δογματικοί σε σχέση με την λεγόμενη δημοσιονομική προσαρμογή, θα πρέπει να μην αγνοούμε την κοινωνική κατάσταση των κοινοτήτων και των χωρών που έχουν φυγεί ιδιαίτερα από τις οικονομικές εξελίξεις. Η κυρία Ριμπέιρο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να χαιρετήσω και εγώ ε, τα πρώτα συμπεράσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Απαιτείται να επιστρέψουμε σε μια περισσότερο βιώσιμη μορφή οικονομικής ανάπτυξης. Θεωρητικά η οικονομική ανάπτυξη πρέπει να λειτουργήσει ευεργετικά για την αγορά εργασίας και για την ανεργία των νέων. Είναι σημαντικό να πάρουν τα κράτη-μέλη μέρος σε μια προσπάθεια αύξησης των ρυθμών ανάπτυξης, αλλά από ό,τι φαίνεται η προσπάθεια αυτή δεν είναι ιδιαίτερα αποδοτική. Απαιτούνται λοιπόν εξελίξεις ε, στον τομέα των επενδύσεων όπως το σχέδιο Juncker. Θα πρέπει επίσης τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν δημοσιονομικές πολιτικές κυρίαρχα υπεύθυνε λαμβάνοντας υπόψη και τις κοινωνικές ανάγκες στα πλαίσια βέβαια της οικονομίας της αγοράς αλλά με συγκεκριμένες κοινωνικές ανησυχίες. Νομίζω λοιπόν ότι με μια αποτελεσματική μορφή τέτοια υπεύθυνη κοινωνικά ανάπτυξης τότε θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε και το πρόβλημα των υπερβολικών ελλημάτων. Τώρα, σχετικά με την βιωσιμότητα των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, οι απειλές είναι πάρα πολύ συγκεκριμένες, τίθεται και θέμα επικουρικότητας. Γνωρίζουμε ότι στον τομέα των συνταξιοδοτικό, στον τομέα των επιδετήσεων στην ανεργία, υπάρχουν εθνικά χαρακτηριστικά που διαφοροποιούν την κατάσταση και που επηρεάζουν την βιωσιμότητα των συστημάτων αυτών. Σε ποιο βαθμό τώρα γίνεται υπόψη αυτή η διαφορά και σε ποιο βαθμό ε, χρησιμοποιούνται τα ειδικά χαρακτηριστικά. Το θέμα δεν είναι να κάνουμε μόνο ε, με γραπτό τρόπο συστάσεις και να καθορίζουμε συγκεκριμένα ποσά. Το θέμα είναι να αναγνωρίσουμε τις προσπάθειες που κάνουν οι Ευρωπαίοι, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και γι' αυτό απαιτείται και τα ευρωπαϊκά όργανα να έχουν μία φωνή. Δεν μπορούμε από τη μία να συγχαίρουμε τους πολίτες για τις προσπάθειες τις οποίες κάνουν και από την άλλη να λέμε ότι μένουν πάρα πολλά ακόμα να κάνουν και η κατάσταση δεν έχει βελτιωθεί. Η κυρία Μάκιντάερ. Thank you. Σας ευχαριστώ. Χαιρόμαστε που βλέπουμε ότι είναι θετική η εκτίμηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Ηνωμένο Βασίλειο, όπου αναφέρεται ότι η οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται, ότι συνεχίζει να πέφτει η ανεργία και ότι η απασχόληση αναμένεται να συνεχίσει να αναπτύσσεται με γοργούς ε, ρυθμούς. 1,9% με λόγια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οι τελευταίες μελέτες της περασμένης εβδομάδας επιβαίνουν αυτή την τάση. Αύξηση λοιπόν αποσχολησιμότητας, 2 εκατομμύρια άτομα παραπάνω σε θέσεις εργασίας σε σχέση με το παρελθόν και αριθμός έκπληξη ε, πολλές γυναίκες ε, στην αγορά εργασίας. Τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι οι διαστατικές μεταρρυθμίσεις είχαν θετικό αντίκτυπο στο επίπεδο αποσχολησιμότητας και τον περασμένο μήνα το συμπεράσματα του Συμβουλίου ΙΚΟΦΗΝ διευκρινίσαν ότι χρειάζονται μεγάλη δέσμευση για διαστατικές μεταρρυθμίσεις σε όλα τα κράτη-μέλη συμπεριλαμβανομένων και των σωστών όρων για την ανάπτυξη και για τη θέση απασχόληση. Κοιτώντα λοιπόν τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να βοηθήσει τα κράτη-μέλη, θα συμφωνούσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι μειώνοντα την περιπλοκότητα τη νομοθεσία μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα σωστό πλαίσιο για τι επιχειρήσει για να δημιουργούν θέσει απασχόληση. Και συγκεκριμένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πιστεύει ότι μειώνοντα την περιπλοκότητα κάποιων συγκεκριμένων νομοθετημάτων μπορούμε να προωθήσουμε την αλλαγή και να αναθεωρήσουμε και να μεταρρυθμίσουμε σε βάθος χρόνου την αγορά εργασίας. Για παράδειγμα, 16 από τα 20 κράτη-μέλη χρησιμοποιούν opt-out για, τα, για τις ε, χρόνους απασχόλησης. Μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι θα πρέπει αυτό το νομοθέτημα να αποσυρθεί για να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη να δημιουργούν πιο πολλές και πιο σωστές θέσεις εργασίας. Ευχαριστώ πολύ, λέει Πρόεδρος. Ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης θα ήθελε να πάρει το λόγο για να απαντήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις σας. Για την πρώτη ερώτηση. Για την οικονομική ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ευρωζώνη. Βλέπουμε ότι ενισχύεται σταδιακά έχουμε κάπως πιο θετικά στοιχεία στις προβλέψεις τώρα από ότι το χειμώνα. Συνεπώς, ο δικός μας στόχος είναι να ενισχύσουμε την ανάκαμψη αυτή. Και πιστεύω ότι το μείγμα πολιτικών, νομισματική δηλαδή με ουδέτερη φορολογική, γιατί ελπίζουμε σε κάτι καλύτερο φέτος, είναι το πιο αποτελεσματικό μείγμα πολιτικής στη σημερινή κατάσταση. Είναι όμως αλήθεια ότι η ανάπτυξη στηρίζεται από κάποιους βραχυπρόθεσμους παράγοντες. Ε, χαμηλές ε, τιμές στο πετρέλαιο, την οικονομική χαλάρωση που αντιστοιχεί σε ένα πιο δύναμο ευρώ επίσης δεν θα τους έχουμε αυτούς τους παράγοντες για πάντα, οπότε πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αυτή την εποχή σωστά, με σοφό τρόπο, ώστε να αντιμετωπίσουμε τα διαφορετικά ζητήματα στις οικονομίες μας. Στη συνέχεια, για τις ερωτήσεις σας όσον αφορά την ε, ανεργία των νέων. Η απασχόληση των νέων είναι προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θέλουμε πραγματικά να εφαρμόσουμε την πρωτοβουλία αυτή για τους νέους που ανακοινώθηκε πρόσφατα και προωθούμε χρηματοδότηση για τις χώρες μέλη που υποφελούνται από την εγγύηση για τους νέους. Και ελπίζουμε οι χώρες μέλη να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια αυτά όσο γίνεται πιο γρήγορα. Και κάποια στοιχεία στις εκθέσεις μας για να επανέλθω στην προηγούμενη ερώτηση υπάρχει το στοιχείο της σύγκλησης, σύγκληση μεταξύ χωρών μελών, αλλά και σύγκληση μέσα στις χώρες μέλη. Σίγουρα είναι προτεραιότητα και για μας να μην υπάρχουν διαφορές μέσα στις χώρες. Συζητάμε επίσης και την ιδέα ε, οροφών, ορίων για την κοινωνική προστασία. Για την επίδοση του Ηνωμένου Βασιλείου, ναι, είναι αρκετά καλές οι επιδόσεις. Όσον αφορά την πολυπλοκότητα των ρυθμίσεων, ξέρετε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόσφατα άρχισε ε, το, την πρωτοβουλία που ονομάζεται ε, καλύτερη νομοθεσία με την πρωτοβουλία REFIT που ακριβώς αυτό το σκοπό έχει η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση να είναι πιο αποτελεσματική Ίσως ε, οι συνάδελφοι να μπορούν να πούν περισσότερες λεπτομέρειες πάνω σε αυτά. Ευχαριστούμε, Μαρία Τάισεν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για να πω στον κύριο Σάντ πρώτα απ' όλα. Να επαναλέβω και εγώ αυτά που είπε και ο κύριος Βάλτης, ο Βάλτης πριν από λίγο. Βάλτης τον Πρόφσκης. Ναι, θέλουμε να έχουμε ένα ελάχιστο επίπεδο κοινωνικής προστασίας και περισσότερη σύγκληση και μεταξύ των χωρών μελών και μέσα στις χώρες μέλη. Αυτό το επαναλαμβάνω κι εγώ. Και σας ενθαρρύνω να μας στηρίξετε και να στηρίξετε την έκθεση των πέντε προέδρων και του Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του ίδιου, και να υπάρξει συμφωνία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να μπορέσουμε πράγματι να βαθύνουμε περισσότερο στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση, γιατί είναι η κατεύθυνση στην οποία όλοι θέλουμε να πάμε. Προς την κυρία Ριμπέιρο. Πώς μπορούμε να καταστήσουμε τα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης περισσότερο βιώσιμα. Αυτό είναι μια πραγματική πρόκληση. Και αν δείτε τι ειδικέ αναχώρας συστάσεις είναι κάτι που και εμείς θέλουμε να ενθαρρύνουμε. Θέλουμε να ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη. Και γι' αυτό, επειδή δεν είναι μόνο στα χέρια τους, θέλουμε να τους δώσουμε συστάσεις για να βελτιωθεί το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης. Και οι συστάσεις μας, οι ειδικές συστάσεις, έχουν να κάνουν και με αυτό. Γιατί είναι σημαντικό για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση το ασφαλιστικό σύστημα. Και ο λόγος που τονίζουμε τόσο πολύ και για την υγεία και για τις συντάξεις την αποτελεσματικότητα τη σχέση κόστους ωφέλους, γιατί πολλά πράγματα μπορείς να βελτιώσεις για να βελτιώσεις την πρόσβαση στην υγεία. Οπότε πάνε μαζί βιωσιμότητα στα συντοξιδητικά και πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Οι συντάξεις να είναι κατάλληλες. Και προς την κυρία Μάκεντάιρ θέλω να πω ότι φυσικά και χρειαζόμαστε καλύτερη νομοθεσία, όχι λιγότερη, το λιγότερη περισσότερη δεν λέει πολλά. Γιατί εξαρτάται από την ποιότητα της νομοθεσίας. Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι καλύτερη νομοθεσία. Γι' αυτό και υπάρχει αυτό το πακέτο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θέλουμε να δούμε δηλαδή πώς μπορούμε να βελτιώσουμε την νομοθετική ρύθμιση σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ελπίζουμε ότι και οι χώρες μέλη θα ακολουθήσουν. Εδώ θέλω επίσης να αναφερθώ και στο πακέτο μεταρρυθμίσεων. Και, συγγνώμη, ε, επενδύσεων, επενδύσεων. Μιλάμε για το ταμείο αυτό, αλλά συγχρόνως θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον, ένα καλύτερο κλίμα για να έρθουν επενδύσεις και επενδύσεις να ανθίσουν. Θέλουμε να βελτιώσουμε συνεπώς και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Είναι στην ημερήσια διάταξή μας γιατί θέλουμε να είμαστε πιο ανταγωνιστικοί και να δώσουμε ευκαιρίες στις επιχειρήσεις να πάνε καλύτερα διασφαλίζοντας όμως κοινωνικές συνθήκες. Και εδώ υπάρχει περιθώριο για βελτίωση σίγουρα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μοσκοβισή τώρα. Σύντομα θα επανέλθω σε αυτά τα οποία έλεγε η προηγούμενη ομιλήτρια για τη σχέση ανάμεσα στη συγκυρία και τις μεταρρυθμίσεις. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο οικονομικής ανάπτυξης, ανάκαμψης, αδιαμφισβήτητο είναι αυτό Πρόκειται για μια κυκλική ανάκαμψη η οποία πιέζεται από ευνοϊκούς ανέμους που γνωρίζουμε, ε, χαμηλό κόστος ενέργειας, ε, χαμηλά επιτόκια, χαμηλός ε, πληθωρισμός και αύξηση αποδοτικότητας. Έχουμε λοιπόν κάθε λόγο να πιστεύουμε με κάποιες επιφυλάξεις βέβαια εφόσον λύσουμε και κάποια θέματα τα οποία έχουμε τα δεδομένα αυτά είναι ισχυρά μεν, κυκλικά δε. Αυτό σημαίνει ότι σε μία κάποια φάση η κυκλική αυτή τάση θα αναστραφεί. Κάθε ευνοϊκός άνομος κάποια στιγμή θα, θα φυσήξει και ανάποδα. Συνεπώς λοιπόν θα πρέπει να προσπαθήσουμε να ενισχύσουμε την οικονομία μας και με διαφορετικό τρόπο η ε, πραγματική ανάπτυξη είναι πολύ χαμηλή, είναι γύρω στο 1%. Πρέπει λοιπόν να καταστήσουμε τον ρυθμό αυτό ισχυρότερο και το τρίπτυχο της Επιτροπής μας είναι πρώτον δημοσιονομική εξυγίανση που να μην βλάπτει την ανάπτυξη, δεύτερον μεταρρυθμίσεις που να μην φύγουν την απασχόληση και τρίτον επενδύσεις που θα επιτρέψουν να καλύψουμε την δυσκολία που έχουμε, τη μεγαλύτερη πρόκληση της επενδύσεις. Λοιπόν, είμαστε 15% πιο χαμηλά από ό,τι στην αρχή της οικονομικής κρίσης. Γι' αυτό λοιπόν αν συνεχίσουμε με τέτοιο τρόπο τότε θα καταλήξουμε σε 10 χρόνια σε οικονομίες δευτέρου επίπεδου. Δεν πρόκειται να το δεχτούμε λοιπόν αυτό. Πρέπει να δημιουργήσουμε επενδύσεις σε τομείς που θα δημιουργούν με τη σειρά τους απασχόληση. Σας ευχαριστώ και αύριο η Ολομέλεια θα εγκρίνει το σχέδιο Juncker. Θα αποτελέσει λοιπόν ένα βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Να δώσουμε λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία Λούκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα ήθελα να μιλήσω στα γερμανικά και η ερώτησή μου απευθύνεται προς τον κύριο Ντομπρόφσκης. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω για τις δύο χώρες, την Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γαλλία. Και οι δύο έχουν υπερβολικό έλλειμμα άνω του 3% στην περίπτωση της Γαλλίας. Πρόκειται για την τρίτη φορά που γίνεται τέτοια διόρθωση που γίνεται τέτοια αναβολή στη διόρθωση του υπερβολικού ελλείμματος και κάθε φορά να δίνεται 6 χρόνια διάστημα. Μέχρι το 2017 τώρα στις συστάσεις αναχώρα για τη Γαλλία αναφέρεται ότι αυτή η παράταση εξαρτάται αποκλειστικά από το κατά πόσο η Γαλλία θα εισαγάγει αποτελεσματικά μέτρα. Μετά τις 10 Ιουνίου του 2015 θα ελεγχθεί κατά πόσον έχουν επιβληθεί και περάσει αυτά τα μέτρα. Ερωτώ λοιπόν κύριε Επίτροπε, Ποια μέτρα έχουν πραγματικά εφαρμοστεί στην ε, Γαλλία προκειμένου ε, να δικαιολογηθεί αυτή η προσωρινή αναστολή που έχει δοθεί στην ε, Γαλλία για την τήρηση των ορίων για το υπερβολικό έλλειμμα και γιατί στην Ενωμένο Βασίλειο δεν έχουν θεωρηθεί επαρκείς αυτές οι εγγύησεις που δίδονται παρά το γεγονός ότι στον Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν λιγότερες παραβιάσεις των ε, συστάσεων ανά χώρα και των όρων που ορίζονται για το περιβολικό ε, έλλειμμα. Μήπως υπάρχουν διπλά μέτρα και σταθμά. Μήπως οι χώρες που βρίσκονται μέσα στην Ευρωζώνη αντιμετωπίζουν πιο ήπια μεταχείριση από ότι οι χώρες που βρίσκονται εκτός Ευρωζώνης. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πρόεδρος θα κάνουμε ένα γύρο ερωταπαντήσεων. Ο Μίκαλ Τόιρερ από την ομάδα των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε, κύριε Επίτροπε Τάισιν, κύριε Επίτροπε Μοσκοβίση, θα ήθελα εξ ονοματός της ομάδας της ΑΛΔΕ για τα θέματα των συστάσεων ε, αναχώρα να ρωτήσω το εξή. Καταρχά, έχουμε το θέμα του δεσμευτικού χαρακτήρα, του υποχρεωτικού χαρακτήρα. Το ερώτημα του πόσο εφαρμόζονται, σε τι βαθμό εφαρμόζονται οι συστάσεις ανά χώρα. Γιατί συζητήσαμε πολύ για την ε, έλλειψη υποχρεωτικού χαρακτήρα για τις χώρες. Έχετε την εντύπωση λοιπόν τα κράτη-μέλη εντωμεταξύ αντιμετωπίζουν μεγαλύτερη δέσμευση και ενθουσιασμό αυτό το θέμα του ownership, του, της κατοχής αν θέλετε των μέτρων αυτών. Και τι μέτρα χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να το πετύχει αυτό. Δεύτερη ερώτηση. το σύνολο των συστάσεων αναχώρα είναι την εντύπωση ότι υπάρχει ένα συνολικό σχεδιασμό σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ότι αυτός ο συνολικός σχεδιασμός θα μπορούσε να ξεπεράσει τα προβλήματα. Όμως ξέρουμε ότι η ανάπτυξη εξαρτάται από τα προϊόντα τα οποία παράγονται στην αγορά και τα οποία θα πρέπει να έχουν ζήτηση. Για τα προϊόντα θα πρέπει να υπάρχει ζήτηση. Κατά πόσο λοιπόν μπορεί όντω να προκληθεί αυτή η διαδικασία ανάπτυξη και πώς αξιολογείται την τρέχουσα συζήτηση όπου οι ισχυρέ πολιτικές δυνάμεις πιστεύουν ότι με πολιτική επιρροή μπορούν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας ενώ η εμπειρική ουσιαστικά η εμπειρία καταδείκνει ότι αυτές οι κοινωνίες που έχουν μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα είναι οι κοινωνίες που προσαρμόζονται πιο καλά στις παγκόσμιες αγορές. Ο Ευχαριστώ πολύ. Ο ομιλητή, Η κυρία Μαρίν Χάρκιν. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ντομπρόσκε, είπατε ότι πέρασε μία μέρα από τη δημοσίευση της έκθεσης των πέντε προέδρων και πέντε μέρες μετά από μία έκθεση του Κοινωνικού Συμβουλίου των Ηνωμένων Εθνών σε σχέση με τις συμφωνίες σε επίπεδο οικονομικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν επικυρώσει τη σύμβαση αυτή και ε, κάποιες χώρες επίσης όπως και η Ιρλανδία δεν θα μπω σε λεπτομέρειες αλλά λέγεται ότι η απάντηση της Ιρλανδίας ε, στην κρίση συγκεντρώθηκε υπερβολικά στη μείωση των δημοσίων δαπανών και έφυξε την κοινωνική προστασία, την κοινωνική κατοικία, την υγεία κτλ. Δηλαδή τους ιδιαίτερα εύθραυστους ε, ε, τομείς του πληθυσμού. Και λέγεται ε, συγκεκριμένα ότι τα μέτρα λιτότητας πρέπει σταδιακά να ανερεθούν και η εφαρμογή των ρυθμίσεων αυτών που προβλέπουν τα Ηνωμένα Έθνη να, να συνοδεύσει τις προσπάθειες οικονομικής ανάκαμψης της Ιρλανδίας θα πρέπει επίσης ε, να χρησιμοποιηθούν κάποια επιπλέον κέρδη από τις καλύτερες οικονομικές συνθήκες ε, και δυστυχώς δεν υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία στις προτάσεις τις οποίες εσείς κάνετε σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μείωση των μέτρων λιτότητας. Η ερώτησή μου λοιπόν δεν αφορά βέβαια μόνο την Ιρλανδία, ε, εσείς σαν Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνετε υπόψη σας τις ανηλυμένες υποχρεώσεις πολλών κρατών μελών στα πλαίσια της σύμβασης αυτής των Ηνωμένων Εθνών. Επηρεάζεστε από αυτή την Διεθνή Δεσμευτική Συμφωνία και αν ναι πού το δείχνετε αυτό στις προτάσεις τις οποίες κάνετε αναχώρα. Γίγκολντ. Uh, Ευχαριστώ τους επιτρόπους που παρουσίασαν τις απόψεις τους για τις ε, αναχώρα συστάσεις. Ε, δύο βασικά ερωτήσεις παρατηρήσεις. Καταρχάς, οι συστάσεις αυτές ε, περιλαμβάνουν υποτίθεται και μια περιβαλλοντική ε, διάσταση. Δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο όμως. Το 2014 υπήρχαν οκτώ συστάσεις οι οποίες ε, είχαν ακριβώς σαν στόχο το λεγόμενο πρασίνισμα. Υπήρχαν επίσης και τρεις συστάσεις για την μείωση ε, επιδοτήσεων βλαβερών για το περιβάλλον και 17 συστάσεις για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την στροφή στις ανανεώσιμες πηγές. Στις συστάσεις τώρα του 2015 δεν υπάρχει παρά μόνο μία σύσταση ε, σε σχέση με τα θέματα της φορολογίας, καμία σε σχέση με τις βλαβερές επιδοτήσεις και καμία σε σχέση με τα ανανεώσιμα. Δηλαδή η λεγόμενη πράσινη ατζέντα την εξαφανίσατε, παραδοθήκατε, δεν ε, αναφέρεστε καθόλου στο περιβάλλον. Είμαι πολύ απογοητευμένος γι' αυτό. Είναι εναντίον φυσικά η στάση σας των ε, υπεσχημένων από πλευρά σας έχετε χαμηλώσει πάρα πολύ τις οικολογικές ανησυχίες και θέλω να μάθω το γιατί. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι για τους οποίους το πρασίνισμα της οικονομίας οδηγεί και στην ανταγωνιστικότητά της. Γιατί το εξαφανίσατε. Και τέλος, σχετικά με την παρουσίαση της παρακολούθησης αν θέλετε της εφαρμογής των μέτρων αυτών από τα κράτη-μέλη για να μάθετε τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Ε, επαφίεστε στα κείμενα εργασίας. Γιατί να μην υπάρχει ένας πίνακας αποτελεσμάτων συγκρίσιμος ε, έτσι ώστε να βλέπουμε αν τα κράτη-μέλη παίρνουν σοβαρά τις αποφάσεις τους. Ευχαριστώ. Ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόσκης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις σας. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τα υπερβολικά ελλείμματα στον Ηνωμένο βασίλιο τη Γαλλία κλπ. Πρώτον, πρέπει να σημειώσουμε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο εξαιρείται από τις τακτικές διαδικασίες και από τον μηχανισμό ενδεχομένων κυρώσεων. Οπότε στην περίπτωση του Ηνωμένου Βασιλείου, ναι, τι κάνουμε. Βάζουμε το συμπέρασμα ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν ανέλαβε επαρκή δράση προκειμένου να αντιμετωπίσει το υπερβολικό του έλλειμμα, αλλά δεν δίνουμε συνέχεια, δεν προβλέπονται διαδικασίες τέτοιες. Στην περίπτωση της Γαλλίας, η Γαλλία συμμετέχει στον μηχανισμό οικονομικής διακυβέρνησης, οπότε σωστά η Γαλλία έπρεπε να υποβάλει τις προτάσεις της, τις δημοσιονομικές μέχρι τη 10η Ιουνίου, κάτι το οποίο έκανε. Και εδώ θέλω να υπογραμμίσω ότι όταν επεκτείναμε για το 2017 τα μέτρα, ήμασταν σαφείς ότι η Γαλλία πρέπει να προχωρήσει σε περισσότερες διαθετικές μεταρρυθμίσεις και δημοσιονομικά πρέπει να προσαρμοστεί κατά 0,2% του ΕΠ φέτος. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντικατοπτρίζεται και στην απόφαση του Συμβουλίου. Τώρα, όπως είπε και ο Πιέρ, αξιολογούμε την πρόταση της Γαλλίας για να δούμε κατά πόσο συνάδει με τις συστάσεις του Συμβουλίου και την ανάλυση μας θα την έχουμε πολύ γρήγορα. Πάντως είναι σημαντική η διαφορά το ότι εξαιρείται από κάποιες διαδικασίες το Ηνωμένο Βασίλειο, ενώ η Γαλλία όχι. Αυτό όπως καταλαβαίνετε κάτι σημαίνει. Όσον αφορά τώρα την εφαρμογή των συστάσεων και την οικειοποίηση των ε, συστάσεων αυτών. Πώς προσπαθούμε να πιέσουμε για εφαρμογή των συστάσεων. Όντω αυτό σημαίνει ότι οι ίδιες οι χώρες μέλη πρέπει να δεσμευτούν περισσότερο. Μέχρι τώρα έχουμε καταλάβει ότι οι χώρες μέλη αντιλαμβάνονται καλύτερα το μηχανισμό, αντιλαμβάνονται καλύτερα το λόγο των συστάσεών μας και έτσι στο τέλος καταλήγουμε σε πιο ισορροπημένες δράσεις και μέτρα που να μπορούν να δεχτούν οι χώρες μέλη και οι κοινωνίες τους. Για τον ε, κοινό ε, σχεδιασμό έχει να κάνει και με την ενιαία αγορά, με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση, το κοινό νόμισμα, Όλα αυτά σημαίνουν ότι φυσικά και χρειάζεται συντονισμός κάποιων πολιτικών. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνουμε σε αυτό το στάδιο. Έρχομαι τώρα στα έγγραφα του ΟΗΕ και το διεθνό επίπεδο στο οποίο δουλεύουμε. Έχω ήδη υπογράψει ότι θέλουμε να υπογραμμίσουμε την κοινωνική διάσταση. Η ε, κυρία Τέσεν ίσως να μπορέσει να επεκταθεί περισσότερο πάνω σε αυτό. Έρχομαι τώρα στην περιβαλλοντική διάσταση. Όπως είπα και στην ε, εισαγωγή μου, έχουμε μειώσει τον αριθμό των ε, συστάσεων και μεταξύ άλλων έχουμε εφαρμόσει μία αρχή. Δηλαδή προσπαθούμε να μην προχωρήσουμε σε επικάλυψη με άλλες πολιτικές. Και έτσι μπορούμε να συζητήσουμε σε άλλα πολιτικά πλαίσια τα θέματα της ενέργειας, της, ε, του ενεργειακού εφοδιασμού, το θέμα των εκπομπών. Κάποιες ειδικέ συστάσεις προς χώρες ε, μέλη μπορεί να έχουν εξαφανιστεί. Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν συνεχίζει να παρακολουθεί ε, τα πράγματα αυτά στις χώρες μέλη. Και αν δούμε ότι υπάρχουν προβλήματα, καθυστερήσεις, πάντα μπορούμε να επαναφέρουμε τα ζητήματα αυτά. Οι συνάδελφοι τώρα ίσως να έχουν να προσθέσουν. Παρακαλώ. Ναι, θέλω να συμπληρώσω λιγάκι αυτά που ακούσαμε από το Βάλτης. Όσον αφορά τη Γαλλία, Γαλλία Ηνωμένο Βασίλειο και τις διαφορές τους υπάρχει κάτι συγκρίσιμο μεταξύ των δύο αυτών χωρών. Είναι ότι η Γαλλία πήρε νέα προθεσμία προκειμένου να τηρήσει τις υποχρεώσεις της απέναντι στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης 2016-2017. Συνεπώς, η ίδια προθεσμία είναι, τα είπε και ο Βάλτης, για τη Γαλλία είναι τρίτη φορά. Υπάρχουν όμως δύο διαφορές. Η πρώτη είναι, και το γνωρίζουν νομίζω αυτό όλοι, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετέχει στην Ευρωζώνη, δεν είναι μέλος της Ευρωζώνης. Οπότε οι δεσμεύσεις που αναλαμβάνει το Ηνωμένο Βασίλειο θα έλεγα ότι είναι λιγότερο δεσμευτικές, λιγότερο υποχρεωτικές από ό,τι για τη Γαλλία. Και οι συνέπειες των αποφάσεων θα έλεγα ότι είναι λιγότερο, ας μην πω σημαντικές, αλλά λιγότερο δεσμευτικές. Το... Η δεύτερη διαφορά είναι ότι για το Ηνωμένο Βασίλειο έπρεπε να κάνουμε την παρατήρηση ότι δεν υπήρχε αποτελεσματική δράση. Πρόκειται για παλιότερη σύσταση που είχε αρχίσει από το 2009 που έλεγε ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έπρεπε να μειώσει το έλλειμμα κατά 75% ετησίως. Αυτό δεν έγινε και γι' αυτό είπαμε δεν ανελήφθη αποτελεσματική δράση, έπρεπε να το πούμε και στη συνέχεια να δώσουμε νέα προθεσμία. Στην περίπτωση της Γαλλίας η κατάσταση δεν είναι ίδια, γιατί τα τελευταία τρία χρόνια, τρεις τελευταίες προθεσμίες ήταν τέτοιες όπου η Γαλλία δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν είχε αποτελεσματική δράση. Τώρα κοιτάμε τι γίνεται μέσα στο 2015 και αυτό θα κληθούμε να κάνουμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Και αυτή είναι λοιπόν μια διαφορά. Αναφέρετε τις συνθήκες. Ναι, αυτό ακριβώς κάνουμε. Πρόκειται για το Σύμφωνο Ανάπτυξης. Και τη δεύτερη παρατήρηση. Το ownership. Η... Το να νιώθουν κάτω στα μέτρα οι χώρες, ο ανστερνισμός. Είχαμε μιλήσει για στατιστικές που δεν είναι αρκετές. Αλλά όσο οι συστάσεις εκλαμβάνονται σαν συστάσεις απ' έξω, τόσο λιγότερο τηρούνται. Γι' αυτό και λέμε ότι θέλουμε προοδευτικά να βελτιωθεί αυτό. Και όπως υπόθηκε ήδη, Ακούσαμε για το περιβάλλον κάποιες παρατηρήσεις πριν. Δεν εγκαταλείπουμε το περιβάλλον. Υπάρχουν οι συστάσεις της Επιτροπής. Γι' αυτό κάναμε λιγότερες συστάσεις. Λοιπόν, περισσότερες στρατηγικού χαρακτήρα με άνοιγμα. Και γι' αυτό πιστεύουμε ότι είναι χρέος μας να εξηγούμε καλύτερα στα εθνικά κοινοβούλια και στις κοινωνίες και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Γιατί με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι οι συστάσεις μας θα γίνουν περισσότερο κατανοητές και θα τηρηθούν έτσι πολύ πιο εύκολα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Λέει Πέτρος. Ναι, λυπάμαι. Ξέχασα να απαντήσω σε μία ερώτηση για τις ε, πληροφορίες ε, για την εφαρμογή και κατά πόσον είναι εύκολη, στην ε, ερμηνεία τους και σε διαφορετικούς πίνακες υπάρχουν πίνακες εύκολοι προς την ερμηνεία. Τέτοιες ε, εκθέσεις για τις συστάσεις ανά χώρα και που περιλαμβάνουν και τι πρόοδος έχει γίνει. Ε, λίγη πρόοδος, μεγάλη πρόοδος, ε, πλήρης εφαρμογή. Υπάρχουν ακόμα και εικόνες. Άρα υπάρχουν πίνακες, weather reports ονομάζονται, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εύκολη κατανόηση. Ερώτηση. Κάναμε την ανάλαση, αλλά δεν υπάρχει συγκριτικός πίνακας για όλα τα κρατημέλη που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί εύκολα για να ασκηθεί πίεση στα κρατημέλη για να εφαρμόσουν. Αυτός ο πίνακας είναι τεχνικός, φαίνεται τεχνικός και προφανώς γι' αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι και είναι κρίμα. Θα ήταν πιο εύκολο να ασκήσει τα μεγαλύτερη πίεση στα κρατημέλη. Θα προσπαθήσουμε, λέει ο κ. Δομπρόσκης, αλλά εκτός μικροφώνου δυστυχώς. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα συγκριτικό πίνακα μεταξύ των κρατών μελών. Αυτό είναι πραγματικά εφικτό και προφανώς είναι προς το συμφέρον μας να υπάρχει μια απεικόνηση απλή και εύκολη του τι συμβαίνει σε κάθε κράτος μέλος αλλά και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος. Ε, η κυρία Τάισεν θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, θα είμαι πάρα πολύ σύντομη για την ερώτηση της κυρίας Χάρκιν. Φυσικά λάβαμε υπόψη τις διεθνείς υποχρεώσεις και τις δικές μας υποχρεώσεις στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στις συμφωνίες που έχουμε συνάψει, αλλά θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και προηγούμενη πραγματικότητα. Η πραγματικότητα λοιπόν τι υπαγορεύει. Ότι πρέπει να εργαστούμε σε τρία μέτωπα. Εξακολουθούμε να έχουμε χρηματοοικονομικά προβλήματα, εδώ θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε. Έχουμε προβλήματα στην παρούσα φάση αλλά έχουμε και τον αέρα στα πανιά μα, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Κατά δεύτερον, θα πρέπει να κάνουμε διαδικαστικέ μεταρρυθμίσει για να φροντίσουμε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη βιωσιμότητα. Προκειμένου και στο μέλλον να υπάρχει μια πιο βιώσιμη κατάσταση. Αυτό προσπάθησαν να το πατήχουν και η προηγούμενη Επιτροπή και το προηγούμενο Κοινοβούλιο. Ξέρουμε ότι χρειαζόμαστε πιο πολλέ επενδύσει, ότι έχουμε το πακέτο των επενδυτικών σήμερα. Και Κατά τρίτον, ε, στο πακέτο της ετήσιας ανάπτυξης, ε, όπου ξεκινήσαμε πέρσι τις εργασίες μας, τότε τις συστάσεις αναχώρα, για τις διάφορες χώρες, κυρία Χάρκιν, θα διαπιστώσετε ότι για μια σειρά χωρών, μεταξύ των οποίων και τη Ιρλανδία, έχουν γίνει συστάσεις προκειμένου να πετύχουμε κάτι παραπάνω για τη συμπερίληψη των πιο ευάλωτων ομάδων ανθρώπων, να δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία στα άτομα αυτά. Και προκειμένου η ανάπτυξη να περιλαμβάνει και αυτά τα άτομα για να μην μείνουν πίσω. Ευχαριστώ. Ο πρόεδρο, ευχαριστώ. Ο Πάτρικ Τιλιαρίκ. Ευχαριστώ κυρία και κύριοι Επίτροποι. Σας ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας, αλλά εκπλήζομαι από ένα πράγμα. Ανεξαρτήτως της κατάστασης, από ό,τι ακούω έρχονται πάντα οι ίδιες συστάσεις. Και με ενιαίο, ομοιόμορφο τρόπο, κατά της αγοράς εργασίας, υπέρ της προσωρινότητας της εργασίας, υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, υπέρ της πίεσης των μισθών και άκουσα τον Επίτροπο κύριο Μοσκοβισή να μας λέει το εξής, ότι χθε δεν είχαμε ανάπτυξη και ήταν απαραίτητε οι συστάσεις αυτές, η λιτότητα ήταν απαραίτητη, τώρα υπάρχει ανάπτυξη και θα πρέπει να ενισχύσουμε ακόμα αυτούς τους κανόνες. Κάτι δεν πάει, κάτι δεν καθόλου καλά. Δεν μιλάμε για, τις, για τα τεράστια κέρδη των μεγάλων διεθνών επιχειρήσεων και των τραπεζών δεν μιλάμε ποτέ για κάποια κίνητρα προς τις τράπεζες να δημιουργήσουν και άλλες πιστοτικές δραστηριότητες υπέρ των παραγωγικών επενδύσεων και της απασχόλησης. Μιλάμε για την έκθεση των πέντε προέδρων. Ακριβώς αυτό τον προσανατολισμό ακολουθεί και η συγκεκριμένη έκθεση. Δεν χρειάζεται να δώσω λεπτομέρειες. Πριν γίνει μια τέτοια έκθεση και τελειώνω κύριε Πρόεδρε, εμείς από την αρχή ε, δεν έχουμε παρά μόνο μία φορά τη δυνατότητα να πάρουμε το λόγο. Πριν γίνει μια τέτοια έκθεση, γιατί δεν έγινε πρώτα ένας απολογισμός της εφαρμογής των προηγούμενων συστάσεων τα τελευταία χρόνια από πλευράς του λαού, όχι από πλευράς μακροοικονομικής, από πλευράς των λαϊκών αναγκών. Αντί να, μιλά, μας μιλάτε συνέχεια για μια ενίσχυση της νομισματικής ένωσης, Πότε θα μας μιλήσετε για μια δημοκρατική, οικολογική και λαϊκή ένωση. Καρή Μαντελή. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Έχω μια σύντομη ερώτηση. Δεν δουλεύει το μικρόφωνο σας, πρέπει να αλλάξετε μικρόφωνο κυρία Αντελή; Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι Επίτροποι, έχετε απαρνηθεί τους στόχους μείωσης της ένδυας που καθορίστηκαν στα πλαίσια της στρατηγικής 2020. Αν πράγματι ισχύει κάτι τέτοιο, εγώ θα ήθελα να εκφράσω τον θυμό μου, την οργή μου Κυρίες και κύριοι η Επίτροποι, τι σκοπεύετε εν πάση περιπτώσει να κάνετε για την καταπολέμηση της φτώχειας και την μείωση των ανισοτήτων σε χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο. Εκρήγνεται ο αριθμός των αστέγων, εκρήγνεται ο αριθμός των ανέργων και εκρήγνεται και ο αριθμός αυτών που μένουν σε ακατάλληλη κατοικία. Τι μπορείτε να μας πείτε για να μας διαβεβαιώσετε για το κοινωνικό περιεχόμενο των προτάσεών σας. Εμείς ανησυχούμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει μια πραγματική έλλειψη καθαρά κοινωνικών προτάσεων. Ζητάμε εδώ και πολλά χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ε, κάποια ελάχιστα κοινωνικά επίπεδα, ένα ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα, μια ατζέντα για τις πράσινες δουλειές απασχόλησης, ε, Πράσινες θέσεις απασχόλησης. Ξέρετε ότι ο 21ος αιώνας υποχρεωτικά θα είναι ένας αιώνας μεταβατικός στον τομέα της ενέργειας και το μέλλον ακριβώς των πράσινων θέσεων απασχόλησης είναι ε, και στα χέρια σας. Λοιπόν, τι θα κάνετε έτσι ώστε τέτοιου είδους ανησυχίες να ληφθούν σοβαρά υπόψη. Κύριε Μοσχοβησή, ήσασταν υπουργό Οικονομικών στην Γαλλία. Κοιτάξτε, μιλάτε πάρα πολύ ώρα. Ε, είχατε πει ότι θα δημιουργήσετε ένα ταμείο αποζημίωσης για τους ανέργους. Κοιτάξτε, σας παρακαλώ σεβαστείτε το χρόνο σας, γιατί αλλιώς δεν θα μπορέσουν να μιλήσουν οι επόμενοι προγραμματισμένοι ομιλητές και κανείς άλλος δεν θα πάρει το λόγο. 1,5 λεπτό, μπορεί να είμαι λίγο ανεκτικός, όχι όμως πάνω από δύο λεπτά. Η κυρία Ματίας έχει το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπη για την παρουσία σας εδώ σήμερα. Μία παρατήρηση. Κάθε φορά που μιλάμε για το λεγόμενο ownership, την αίσθηση του ανήκειν ή τη συμμετοχή στις προτάσεις αυτές, ακούγεται λίγο αστείο, λίγο περίεργο. Ε, ταυτόχρονα με αυτή την πρόταση το μόνο που κάνετε είναι να απειλείτε και να εκβιάζετε τα κράτη-μέλη πάνω στα μέτρα τα οποία θα πρέπει να εφαρμόσουν. Κοιτάξτε τι γίνεται στην Ελλάδα στην παρούσα φάση και τι έχει γίνει και σε άλλες χώρες. Εξετάζοντας τις συστάσεις αυτές μου έρχεται και κάτι άλλο στο νου και το οποίο μου φαίνεται σημαντικό. Αντί να λύσουμε τα προβλήματα, η Επιτροπή προτείνει να εφαρμόσουμε πάντα τις ίδιες ε, συνταγές ανεξαρτήτως των αποτελεσμάτων του παρελθόντος. Αντί να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις, ε, δημιουργούμε καινούργια θέματα. Το θέμα το οποίο δημιουργείται τώρα είναι το θέμα της αηφορίας, ε, της βιωσιμότητας μάλλον, των εθνικών συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Το πρόβλημα το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε σήμερα είναι η ανεργία. Αυτό είναι το βασικό θέμα. Τα προβλήματα λοιπόν απασχόλησης στην Πορτογαλία δημιουργήθηκαν από τα προγράμματα προσαρμογής. Χάσαμε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. 300.000 Πορτογάλοι εγκατέλειψαν τη χώρα τους λόγω της λιτότητας αν ήταν στην Πορτογαλία δεν θα είχαν δημιουργήσει προβλήματα στην κοινωνική ασφάλιση. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσετε να λύνετε τα πραγματικά προβλήματα και πώς θα σταματήσετε να δημιουργείτε νέα. Γιατί ο στόχος δυστυχώς τον οποίο έχετε δεν αλλάζει με τίποτα. Και μπροστά στη διάλυση των οικονομικών συστημάτων των κρατών μελών, οι συστάσεις τις οποίες κάνετε είναι συστάσεις μακροοικονομικής άγνοιας Συνεπώς λοιπόν και θα τελειώσω εδώ. Α, κοιτάξτε τελειώνω αφήστε με λέει η κυρία Ματίας. Είναι η τελευταία μου φράση μην με κόβετε. Ετζέα. Ευχαριστώ πρόεδρε. Κύριε Επίτροπη, τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Μιλάτε για δημοσιονομική εξυγίανση, ακόμα και στις συστάσεις αναχώρα. Μιλάτε για ενίσχυση της ανάπτυξης, βάζοντας εμπόδια στην ανάπτυξη. Και επιβάλλετε κυρώσεις αν ε, οι χώρες δεν σεβαστούν ε, ε, τους κανόνες σας. Αυτό το οποίο κάνετε είναι κάτι το οποίο μοιάζει με μια μανιοκαταθλιπτική σχιζοφρενική κατάσταση στην ουσία κάνετε ένα βήμα μπρος και ένα βήμα πίσω, τη μία λέτε το α και στη συνέχεια αναιρείτε το ίδιο το α. Σας εκτιμώ προσωπικά. Αλλά όταν σας ακούω ε, να λέτε ότι θα μπορέσουμε να αναπνεύσουμε τώρα, διότι πράγματι έπεσε συγκεκριμένα η ανεργία κατά 1 ή 1,5%. Για, σκεφτείτε λίγο για πόσους μιλάτε, πόσοι είναι σήμερα στην Ευρώπη οι οποία ζουν με μη ανθρώπινο τρόπο. Πότε εσείς οι επίτροποι θα συνειδητοποιήσετε ότι η χώρα μας και η Ευρώπη έχει ανάγκη από μια βαθιά διαρθρωτική αλλαγή, την προστασία των κοινωνικών συστημάτων. Σας ε, είναι εντελώς ξένο, σας ακούω να αναφέρετε το επίθετο κοινωνικός, αλλά δεν αναφέρεστε στην προστασία των πολιτών. Δεν έχω ακούσει ποτέ τον τελευταίο καιρό προτάσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που να σέβονται την αξιοπρέπεια του πολίτη. Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα θα ακούσουμε και τις επόμενες ερωτήσεις του επόμενου γύρου μαζί, γιατί τελειώς δεν θα προλάβουμε. και οι επίτροποι σίγουρα θα μπορέσουν να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις μαζί. Περνάμε στον πέπτο γύρο. Φαντακεντελάρε. Ευχαριστώ πρόεδρε. Βέβαια όσο πιο αργά παίρνουμε το λόγο τόσο πιο λίγο μπορούμε να μιλήσουμε. Λοιπόν κύριε επίτροπε η μεγαλύτερη πρόκληση σίγουρα είναι η ανεργία σήμερα. Και εκεί όπου υπάρχουν ειδικέ συστάσεις η ανεργία είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει πια σαν κύρια προτεραιότητα την ανεργία, γιατί τη βλέπουμε λιγότερο στις ειδικέ συστάσεις. Αναρωτιέμαι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι θα κάνει γι' αυτό. Thank you, Thomas. Ευχαριστούμε, Τόμας Μαν. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι αυτή η πρώτη ανταλλαγή ήταν πάρα πολύ σημαντική για να ξεκαθαρίσουμε ότι πρόκειται για συστάσεις από χώρα, για δυνατότητες δηλαδή προτάσεων, όχι για επιταγές. Ε, υπάρχει επικουρικότητα η οποία και δεν υπάρχει πρόβλημα λοιπόν. Και μπορούμε να πούμε ότι κάποια στιγμή στο name and shame θα υπάρχει πιο λίγο shame. Αναπτύξουμε λοιπόν το καλό παράδειγμα. Πολύ καλό θα ήταν αυτό. Προς την κυρία Τάισεν, όταν λέμε ότι μία από τις ανάγκες είναι να αναθεωρήσουμε την αγορά εργασίας. Υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι αυτό που υπάρχει στα κράτη-μέλη ε, σε ό,τι αφορά την απορρίθμιση αμφισβητείται. Πώς μπορούμε λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο και δεύτερον τα κονδύλια που έχουμε κατά πόσον είναι ε, ευέλικτα. Όταν διαπιστώνουμε για παράδειγμα ότι στην ε, πρωτοβουλία για την νεολαία προκύπτουν πολύ μικρά κονδύλια στα κράτη-μέλη και δεν υπάρχει δυνατότητα συμμετοχή κάποιων κρατών μελών. Υπάρχει δυνατότητα να δράσουμε κατά προτεραιότητα για να αντιμετωπίσουμε τέτοια εντοπισμένα προβλήματα και ύστερα. Υπάρχει συνέχεια αυτή η αντίφαση. Από τη μία έχουμε τη λιτότητα και την εξοικονόμηση και από την άλλη έχουμε τις επενδύσεις που είναι απαραίτητα. Αλλά αυτά τα δύο πάνε χέρι-χέρι, ε, την εξοικονόμηση δεν μπορούμε να κάνουμε επενδύσεις για να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πώς λοιπόν είσαστε διδεθειμένοι να υποστηρίξετε και να προβάλλετε από επικοινωνιακή άποψη αυτή την ισορροπία που χρειάζεται. Ευχαριστώ. Άνεμανς. Το μικρόφωνο σας. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί οι συστάσει αναχώρα είναι κάτι το οποίο εξετάζουμε συχνά πυκνά για να δούμε τι γίνεται με τι ανισορροπίε αυτέ τι μακροοικονομικέ. Θα πρέπει λοιπόν να αλλάξει κάτι στην προσέγγιση, γιατί αυτή η ανισορροπία είναι ε, εξορισμού κάτι αρνητικό και θα πρέπει λοιπόν να δούμε τις κακές αυτές πολιτικές. Και η Γερμανία λοιπόν ε, ως οικονομικός ε, ε, φορέας πολύ δυνατός, τα πηγαίνει καλύτερα σε ό,τι αφορά ε, τη βαθμολογία στον έλεγχο σε σχέση με το Βέλγιο. Είναι λοιπόν γελίο το γεγονός ότι θα πρέπει να λάβει τέτοιες ε, αποφασιστικές δράσεις η Γερμανία ενώ το Βέλγιο με την νοτιοευρωπαϊκό του χρέος ουσιαστικά θα πρέπει να υποστεί μόνο κάποιες περιορισμένες συστάσεις και ένα περιορισμένο έλεγχο. Ε, ρωτώ λοιπόν, η βελγική κυβέρνηση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τι μέτρα έχει λάβει προσφάτως και ποιος είναι ο μακροοικονομικός αντίκτυπός τους και κυρία Επιτροπή τι θέλετε να κάνετε στο Βέλγιο συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων. Ποια είναι λοιπόν η στόχη με βάση των θα σας κρίνουμε με άλλα λόγια. Ευχαριστώ κύριος Μπάλας. Ευχαριστώ. Ε, για τις διαφορετικές μορφές ανάπτυξης αναφερθήκατε, τα διαφορετικά μέτρα μάλλον για την ανάπτυξη, ε, μείωση της φορολογικής πίεσης στις επιχειρήσεις, αύξηση των επενδύσεων για τις τοπικές και κοινωνικές αρχές, ε, αυτά τα οποία είναι γνωστά. Αλλά δεν μιλάμε για ένα άλλο θέμα σημαντικό το θέμα των στρατιωτικών δαπανών σαν παράδειγμα. Το θέμα της ε, δημογραφίας. De Δεν μιλάμε επίσης για τη μείωση των ε, σχολικών δαπανών. Δεν μιλάμε για τις ανισότητες που αυξάνονται στην Ευρώπη. Ένα θέμα που έχει τεθεί και από το Δέλτα Νιτάφ και από τον ΟΣΑ. Συγγνώμη. Συνεπώς, δεν μιλάμε για την καινοτομία, για την οικολογική μετάβαση και ξέρουμε ότι αυτό είναι βασικό ενδογενές όπλο για την ανάπτυξη. Φοβάμαι ότι κάνουμε λάθος. Μήπως θα πρέπει να αλλάξετε μουσική κύριε Επίτροπη. Εν μόνο για το ΚΑΤΣΤΙΑΙ, η κυρία Σάντερ. Merci, Monsieur le Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κυρία Κύριε Επίτροπε, είναι αλήθεια ότι η οικονομική συγκυρία σήμερα είναι πιο ευνοϊκή και ότι πολύ δειλά επανέρχεται η ανάπτυξη, ακόμα και αν είναι πολύ χαλαρή ακόμα, όπως είπε και ο Επίτροπος Δομπρόφσκι. Η ανάκαμψη αυτή έχει όμως επιπτώσεις διαφορετικές στις διάφορες ευρωπαϊκές χώρες υπάρχουν διαφορετικές επιπτώσεις ανάλογα επίσης με την κατηγορία ανέργων. Το είπαμε αυτό. Υπάρχει κάποια κατηγορία ανέργων που δεν αποφελείται τελικά από αυτή την ανάκαμψη. Πρόκειται για τους μακροχρόνια άνεργους. Είναι το ίδιο αυτό σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Εξού και ερώτησή μου τι πρωτοβουλίες προβλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι χρηματοδότηση, αν υπάρχει τέτοια πρωτοβουλία, τι χρηματοδότηση προβλέπεται για να καταπολεμηθεί η μακροχρόνια ακριβώς ανεργία. Ευχαριστούμε. Ο Αντιπρόεδρος Ντομπρόφσκης πρώτα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω στις ερωτήσεις συνολικά οι περισσότερες πήγαιναν προς την ίδια κατεύθυνση. Πρώτα απ' όλα για την κοινωνική προστασία, την κοινωνική ένωση, πράγματα που έθιξαν διάφοροι ευρωβουλευτές. Σας είπα τι δουλειά κάνουμε φέτος, ότι θέλουμε να ενισχύσουμε την κοινωνική διάσταση του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε πλήρως τους δείκτες για την ανεργία στο Ευρωπαϊκό αυτό εξάμεινο και ανέφερα και την έκθεση των πέντε πρόεδρων που μιλάει για σύγκληση μεταξύ των χωρών μελών αλλά και μέσα στην κάθε χώρα μέλος. Και αυτό για να αντιμετωπιστεί η ένδια. Και μιλήσαμε και για την ε, κοινωνική προστασία που είναι μια νέα ιδέα τώρα στα πλαίσια του εξαμήνου αυτό. Οι πέντε πρόεδροι είναι σαφείς από αυτού. Για αυτήν ε, την έκθεση όμως δεν θα συμφωνήσω με την διατύπωσή σας ότι εσείς ε, καταρτήσατε αυτήν την έκθεση. Όχι, είναι οι πέντε πρόεδροι που εκπώνησαν την έκθεση αυτή. Δεν είμαστε εμείς. Πρόκειται για ένα κοινό έργο των πέντε θεσμικών οργάνων. Μιλήσατε πολύ για την ανεργία. Πράγματι, η ανεργία είναι μία από τις κύριες ανησυχίες μας. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε την ανεργία λοιπόν, διευκολύνοντας πρώτα απ' όλα την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση, αλλά και μέτρα προστασίας, κατάρτισης των ανέργων, διαβίου κατάρτιση έτσι ώστε ο κόσμος να διαθέτει τα προσόντα τα οποία χρειάζονται στην αγορά εργασίας. Επικεντρωνόμαστε λοιπόν στην εφαρμογή του μέτρου υπέρ της νεολαίας, απασχόληση και νεολαία. Αλλά σίγουρα η Ματάισον θα πει περισσότερα. Ρωτήσατε επίσης για διάφορες χώρες μέλη και την κατάστασή τους σε σύγκριση με τη Γερμανία. Εγώ δεν βλέπω εδώ πέρα καμία αντίφαση. Οι χώρες μέλη που έχουν κάποια δημοσιονομική άνεση πρέπει να την χρησιμοποιήσουν για να κάνουν επενδύσεις. Και στην διαδικασία μακροχρόνων ισορροπιών έχουμε ένα όριο του 6% πλεόνασμα σε σχέση με το ΕΠ. Αν το υπερβαίνουν, πρέπει να βρουν τρόπο να το μειώσουν. Συνεπώς, η σύστασή μας προς τη Γερμανία είναι να διευκολύνει τις επενδύσεις και να αντιμετωπίσει τη ζήτηση και να χρησιμοποιήσει και τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό χώρο. Και η Γερμανία έχει ήδη ανακοινώσει πρόσφατα διάφορες πρωτοβουλίες προς τη σωστή κατεύθυνση πακέτο επενδύσεων για τα επόμενα τρία χρόνια, επενδύσεις ειδικά στις περιφέρειες, συνεισφορά στο επενδυτικό σχέδιο Juncker, άρα αντιδράει βάσει των συστασιών μας. Θα σταματήσω. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία αυτή που μας δώσατε να έχουμε ανταλλαγή απόψεων και σίγουρα οι συνάδελφοι θα έχουν να προσθέσουν κάποια πράγματα. Πρόεδρος, δεν είχα δει πριν τον κύριο Πορζάνη ότι ήταν στον κατάλογο. Δεν σας βλέπω, βλέπετε είσαστε εκεί πίσω και ζητώ συγγνώμη που το παρέβλεψα. Θα σας δώσω λοιπόν το λόγο, ένα λεπτό όμως το πολύ. Αν έχετε κάτι να ρωτήσετε και θέλετε τώρα, παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε αυτή την ευκαιρία. Ένα τεχνικό ζήτημα θέλω να θέσω. οι στατιστικές για την απασχόληση, μάλλον για την ανεργία, για το Διεθνές Γραφείο Εργασίας και άλλοι, ε, συζητάνε το θέμα κατά πόσο πρέπει να συμπεριλάβουμε κάποιον που δουλεύει μια ώρα τη εβδομάδα ή όχι. Ή ας πούμε έναν Ούγκρο ο οποίο δουλεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς με αυτές τις στατιστικές πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αν θέλουμε να πάρουμε σωστές αποφάσεις. Ευχαριστούμε. Η Επίτροπος Τάισεν. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, Έγιναν διάφορε παρατηρήσει ότι δεν ασχολούμαστε με του ανθρώπου, αλλά ασχολούμαστε με τα συστήματα. Θα ήθελα να επαναλάβω για όσου δεν το έχουν καταλάβει ακόμα, και αυτό προέκυψε και από τι απαντήσει των συναδέλφων, ότι όλη η πολιτική τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει στο επίκεντρο τη τον άνθρωπο. Και όταν μιλάμε για φορολογικέ, διευθυντικέ μεταρρυθμίσει, όταν μιλάμε για επενδύσει, όλα αυτά ω σκοπό έχουν να βελτιωθεί το πλαίσιο στο οποίο ζει ο άνθρωπο και να δοθεί μεγαλύτερη μεγαλύτερες ευκαιρίες για ένα καλό εισόδημα και για καλύτερη κοινωνική προστασία στους ανθρώπους και για καλύτερη κοινωνική κοινωνικές παρουσιάσεις. Ανέφεραν διάφορες συνάδελφοι, διάφορους στόχους τους οποίους θα έπρεπε να πετύχουμε, με κάποιους εκ τους οποίους συμφωνώ, αλλά θα ήθελα να παρατηρήσω ότι εργαζόμαστε σε ένα νομικό πλαίσιο. Έχουμε αρμοδιότητες, αρμοδιότητες έχουν και τα κράτη-μέλη. Δεν μπορούμε να επέμβουμε εκεί που δεν έχουμε αρμετιότητες. Και γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται συνεργασία στα πλαίσια της Ευρώπης του 2020 και θα πρέπει να βρούμε ένα άλλο σύστημα διακυβέρνησης και να προσπαθήσουμε να δώσουμε κίνητρα. Δεν μπορούμε ασφαλώς όμως να τα ρυθμίσουμε όλα από την Ευρώπη. Πολλά θα πρέπει να αποφασιστούν από κοινού με την Ευρώπη. Αυτό ασφαλώς το ξέρετε και εσείς οι ίδιοι. Ασκήθηκε κριτική ότι δίνουμε μεγάλη έμφαση υπερβολική στη βιωσιμότητα του τομέα της κοινωνικής πρόνοιας, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τις συντάξεις ε, και την υγειονομική περίταλψη. Γι' αυτό αναφέρεστε υποφέτω, μιας και αυτό περιλαμβάνεται στη συστάση αναχώρα. Τι είναι όμως ε, βιώσιμο και κατάλληλο. Πρόκειται για θέματα τα οποία θα φέτουν στην, στο επίκεντρο τα ίδια τα κράτη-μέλη. Στο ΕΜΚΟ λοιπόν το τονίσαμε το ζήτημα αυτό και μας ζητήθηκε ρητά να δώσουμε πιο πολύ προσοχή στο θέμα αυτό και νομίζω ότι καλά κάνουν, δίκιο έχουν και θα πρέπει να φροντίσουμε όχι μόνο να υπάρχει κοινωνική ασφάλεια τώρα, αλλά να μπορεί και η μελλοντική γενιά να έχει μια σωστή κοινωνική προστασία και προκειμένου λοιπόν να επιτευχθεί αυτό θα πρέπει να υπάρχει βιωσιμότητα και να υπάρχει επαρκή κάλυψη εδώ, τώρα και στο μέλλον ο Τόμ Κεντελάρε έθεσε το θέμα του ότι δεν δίνεται επαρκής προσοχή στις συστάσεις αναχώρα στην ενεργεία των νέων και τι μπορούμε να κάνουμε στη μακροπρόθεσμη, για τη μακροπρόθεσμη ενεργεία. Μπορεί να δίνεται αυτή η εντύπωση, αλλά δεν στέκει αυτό. Η προχρηματοδότηση για την εγγύηση για τους νέους βλέπουμε ότι φτάνει το 30%. Αυτό είναι άνευ προηγουμένου στην Ευρώπη. Για να φροντίσουμε οι χώρες που έχουν ε, εμπόδια και αντιμετωπίσουν εμπόδια λόγω του προπολογισμού τους να μπορούν και αυτές να συνεχίσουν και να ξεκινήσουν τα προγράμματα αυτά. Μας υποστήριξε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα ήθελα λοιπόν εκ νέου να σας ευχαριστήσω, αλλά αυτό μας απασχολεί ιδιαίτερα η ενεργεία των νέων σε ό,τι αφορά τον την πρόοδο των κρατών μελών για την ε, ανεργία των νέων. Θα συλλέξουμε στοιχεία και δεδομένα φέτος ε, στα κρατημέλη και θα τα αξιολογήσουμε στα πλαίσια του Youth Guarantee του χρόνου. Και αν χρειαστεί θα πρέπει και εσείς ε, να καλέσετε τις κυβερνήσεις σας στις χώρες σας να εργαστούν σκληρά προς την κατεύθυνση αυτή για να χρησιμοποιήσουμε το μακρο, το πολιτές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο. Αν θέλουμε να πετύχουμε κάτι στην ενεργεία των νέων, θα πρέπει να αποδείξουμε ότι αυτά που έχουμε ήδη κάνει αποφέρουν καρπούς. Όχι, δεν είναι ότι ε, ξοδέψαμε απλά χρήματα, αλλά πετύχαμε και συγκεκριμένα αποτελέσματα. Διάφοροι συνάδελφοι έθεσαν τώρα τη διάσταση της μακροπρόθεσμης ανεργίας και το τι σκοπεύουμε να κάνουμε προς την κατεύθυνση αυτή. Είναι πάρα πολύ επιμόνο αυτό το πρόβλημα, ξέρετε. Και Παρά το γεγονός ότι μειώνονται λίγο η ενεργεία στους νέους, δεν είμαστε κανοποιημένοι ασφαλώς με ποσοστά μεταξύ 9 έως 11% γιατί η ενεργεία θα πρέπει να είναι μηδενική. Ούτε έναν άργο δεν θα θέλαμε να, κάνουμε, να έχουμε. Αλλά ιδιαίτερα η μακροπρόθεσμη ενεργεία είναι ένα πολύ επίμονο πρόβλημα η ανεργία των νέων μειώνεται. Αργά μεν, αλλά μειώνεται. Αλλά η με ανεργία δεν μειώνεται. σα ίσα που αυξάνεται ελαφριά σε κάποια κρατημέλη. Κάτι θα πρέπει να κάνουμε λοιπόν προ την κατεύθυνση αυτή. Ελπίζω πριν το καλοκαίρι να μπορέσω να καταθέσω μια πρόταση προ την κατεύθυνση αυτή για ευρωπαϊκά κονδύλια και συστάσει προ τα κρατημέλη για συνολικά πακέτα για την αντιμετώπιση της μακροπρόθεσμης ανεργία. Έτσι συνήθω Υπάρχουν και κοινωνικά προβλήματα, προβλήματα ε, για τη φύλαξη των παιδιών, ε, προβλήματα υγείας που κρύβονται πίσω από τη μακροπροθεσμή ανεργία. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπιστούν με μια εξωτερικευμένη ε, αντιμετώπιση και μια συνολική προσέγγιση. Τέλος, το σχόλιο του Τόμας Μαν. Μιλήσατε για τη μεταρρύθμιση της αγοράς εργασίας, την την πιο ενεργή ε, πολιτική για την αγορά εργασίας και για την μείωση της προστασίας των ατόμων. Όχι. Όμως όλοι θα πρέπει να θερήσουν στις δυνάμεις τους. Θα πρέπει να μπει ένα τέρμα σε, να μπει ένα τέρμα, τέλος στα συστήματα που αφήνουν ε, ε, έξω τους προσβητέρους τους πιο ηλικιωμένους. Όλοι θα πρέπει να μπορούν να μπουν στην αγορά εργασίας και οι πιο νέοι. Αν θέλουμε να καταπολεμήσουμε την τελμάτωση της αγοράς εργασίας θα πρέπει να δούμε τι γίνεται και με τις επισφαλείς θέσεις εργασίας γιατί υπάρχουν άτομα τα οποία είτε δεν έχουν δουλειά είτε βρίσκονται σε μια επισφαλή θέση εργασίας ε, διαρκώς όμως. Θα πρέπει λοιπόν να καταπολεμήσουμε τον κατακαιρματισμό της αγοράς εργασίας προκειμένου να βελτιώσουμε τις συνθήκες για όλα αυτά τα άτομα. Ελπίζω, Πρόεδρε, να ανέφερα όλα αυτά τα οποία μου τέθηκαν ως ερωτήσεις. Α, και τέλος, ε, ποιους, ε, ποιοι είναι τα αριθμητικά στοιχεία, οι στόχοι για το Βέλγιο. Θέλουμε να μειωθεί η ενεργία στο Βέλγιο και σε όλη την Ευρώπη, όσο πιο πολύ μειωθεί τόσο καλύτερα, και κυρίως η ενεργία των νέων, γιατί θέλουμε να δώσουμε ελπίδα στους νέους και να μην μιλάμε για χαμένες γενιές και κάνουμε ό,τι μπορούμε προς την κατεύθυνση αυτή χρησιμοποιούμε όλα τα μέσα που έχουμε, θα πρέπει να δώσουμε κίνητρα στα κράτη-μέλη και με την ευρωπαϊκή πολιτική θα πρέπει να φροντίσουμε για νέε επενδύσει, για πιο πολλέ θέσει απασχόληση. Προκειμένου οι νέοι να μπορούν να έχουν και πάλι αυτή την πρόσβαση στην αγορά εργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ο Πιέρ Μοσκοβίση, λέει ο πρόεδρο. Ίσως τυχαία οι απαντήσεις μου δεν αρκούν για τους Γάλλους συναδέλφους. Να πω λοιπόν και για τον κύριο Ιαρίκ ότι εμείς δεν έχουμε σαν προτεραιότητα τη λιτότητα. καθένας έχει τους δικούς του ορισμούς βέβαια για το ίδιο πράγμα. Αλλά προτεραιότητά μας είναι η στήριξη της ανάπτυξης, ανάπτυξη και απασχόληση. Αυτό συνδέεται με την ίδια τη συγκυρία ε, η προηγούμενη Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε άμεση κρίση μπροστά της με ανάγκη σταθεροποίησης και διάσωσης του ευρώ. Τώρα τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί και η ατζέντα είναι διαφορετική. Θέλουμε την ανάπτυξη. Δεν θέλω να μακρηγορήσω. Δύο παραδείγματα όμως αυτού του οποίου όπως είπατε δεν κάνουμε. Δεν συμφωνώ με την πρότασή σας. Να σας πω το εξής ε, για, τα τεράστια κέρδη των μεγάλων επιχειρήσεων. Εγώ θα επανέλθω για τα θέματα της φορολογίας είμαι υπεύθυνο και αν σας παρουσιάσω τις δράσεις που προτείνω. Θα πρέπει έτσι ώστε οι πολυεθνικές επιχειρήσεις να σταματήσουν να φοροδιαφεύγουν. Δεν το κάνουν όλες βέβαια αλλά συμβαίνει έχουν νομικές υπηρεσίες που τους επιτρέπουν να παίζουν και να επιλέγουν εθνικά φορολογικά συστήματα που είναι γεμάτα τρύπες ευκαιρίας. Θα πρέπει εμείς ε, να καταπολεμήσουμε αυτή τη δράση. Αυτός είναι ο στόχος του προγραμματός μου και νομίζω ότι θα υπάρξει ομοφωνία από πλευρά σας ε, διότι εγώ ε, προσπαθώ σε προσωπικό επίπεδο να κάνουμε ε, μέτρα ε, για την δίκαιη φορολογία και οι επιχειρήσεις από την άλλη να προσπαθούν μέσω των ειδικών ρυθμίσεων να διαφεύγουν. Λοιπόν, δεν θα πρέπει να υπάρχουν επιχειρήσεις που δημιουργούν, που παράγουν και που δεν πληρώνουν ε, φόρους. Πρέπει να πληρώνουν φόρους οι επιχειρήσεις εκεί όπου παράγουν πλούτο. Τώρα για τις επενδύσεις. Το σχέδιο Juncker αυτό έχει σαν στόχο. Ε, φυσικά οι επενδύσεις δεν είναι πανάκια, αλλά παρόλα αυτά είναι ένα σημαντικό βήμα, ένα διαφορετικό βήμα και για τις μικρομεσαίες. Υπάρχει ένα τμήμα το οποίο ε, έχει σαν στόχο ακριβώς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κυρία Ντέλη, αναφέρθηκε σε προηγούμενες ε, αρμοδιότητές μου. Νομίζω ότι το θέμα του ευρώ είναι κάτι το οποίο εξακολουθούμε να το βλέπουμε με τον ίδιο τρόπο. Θα δούμε στην έκθεση των πέντε προέδρων που θα συζητηθεί υπάρχουν ιδέες οι οποίες δείχνουν ότι προσπαθούμε να λειτουργήσουμε με την αρχική ιδέα που είχαμε για το ευρώ. Και ο κύριος Μπαλάς αναφέρθηκε σε διαφορετικές προτεραιότητες. Κοιτάξτε, εμείς έχουμε την πρώτη ύλη μας στα εθνικά μεταρρυθμιστικά σχέδια. Κάνουμε παρατηρήσεις επί τη βάση μεταρρυθμίσεων που προβλέπουν να κάνουν οι διάφορες χώρες μέλη. Δηλαδή στη Γαλλία το γαλλικό σχέδιο το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά. Εγώ έχω αποσυρθεί κατά κάποιο τρόπο από την γαλλική πολιτική ζωή, ανήκα όμως ε, ε, στο πλειοψηφούν κόμμα, αν και τώρα είμαι υποχρεωμένος να λειτουργώ ουδέτερα. Προσπαθούμε όμως να επιλέξουμε τα μέτρα των κυβερνήσεων και στη συγκεκριμένη περίπτωση της γαλλικής κυβέρνησης τα σχολιάζουμε και προτείνουμε βελτιώσεις. Θα ήθελα λοιπόν, λέει ο κύριος Γκολτιέρη, να ευχαριστήσω τον Αντιπρόεδρο Ντρομπόσκης και τους Επιτρόπους Τάισεν και Μοσκοβισή για μια έντονη ζωηρή συζήτηση ανταλλαγή απόψεων με το Κοινοβούλιο. Στην έκθεση των πέντε Προέδρων υπάρχει και η πρόταση εμβάθυνσης της ανταλλαγής απόψεων για το Ευρωπαϊκό Εξάμεινο των επαφών ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και τα άλλα όργανα και αυτό περιλαμβάνεται ίσως και στην προσπάθεια για μια διοργανική συμφωνία με την Επιτροπή. Ελπίζουμε λοιπόν στα πλαίσια της εφαρμογής του εξαμήνου να συμμετέχουμε και εμείς για μια καλύτερη διακυβέρνηση. Πράγματι έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα νέο μίξ πολιτικής το οποίο ε, θέτει σε λειτουργία η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει αρχίσει να αποδίδει σε μία πρώτη αρχική φάση. Υπάρχουν κάποια πρώτα δείγματα ανάπτυξης, δεν αρκούν. Πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε και με το πρόγραμμα Juncker και με τα άλλα θέματα. Και όπως είπε και ο κύριος Ντομπρόσκης, ε, θα πρέπει να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε το λεγόμενο 3α στο κοινωνικό τομέα. Δεν είναι εύκολο αλλά νομίζω ότι με ε, μέσα όπως οι αυτόματοι σταθεροποιητές και με άλλα μέτρα ε, θα πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και στην έκθεση Μπέρες η οποία θα ψηφιστεί αύριο νομίζω ότι μπορούμε να καταστήσουμε την διακυβέρνηση της Ευρωπαϊκής Νομισματικής Ένωσης πιο αποτελεσματική. Σας ευχαριστώ όλους, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Η Επιτροπή μας θα συνεχίσει να συνεδριάζει. Έχουμε άλλα δύο θέματα, λέει η κυρία Ουλφσκόγκ. Σας δίνουμε όμως κάποιο χρόνο. Ε, ήταν καλό που βρέθηκε χρόνος ε, για αυτήν την ακρόαση. Η προσπάθεια συζήτησης της οικονομίας είναι συζήτηση και προσπάθεια για την απασχόληση. Δύο λεπτά διάλειμμα και θα συνεχίσουμε στα επόμενα θέματα.